Να συνεχίσουμε λοιπόν. Επόμενο σημείο στην ημερία διάταξη, πολιτέ ε, πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Τον Ιανουάριο του 2013 η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την παράταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της ρήπανσης ε, από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και να παρακολουθεί την έκταση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, της ρήπανσης που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και ε, φυσικού αερίου και επίσης επέκτηνε και την γεωγραφική κάλυψη για να καλύψει και τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Με την έκθεσή μου λοιπόν σήμερα ε, δεν θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσον είναι καλή ιδέα ε, και κατά πόσον αυτά τα επιπλέον καθήκοντα είναι καλά ή άσχημα. Αυτό που εξετάζουμε μπορεί ο Ευρωπαϊκός αυτός οργανισμός να ε, χρηματοδοτηθεί καταλήλως για να χρηματοδοτήσει και αυτός αυτές τις δραστηριότητες της επιπλέον μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 160 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα αυτό και 154 ε, εκατομμύρια ευρώ ήταν τα υφιστάμενα καθήκοντα συν 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νέα καθήκοντα. Αυτό για να σας ε, ε, πω λίγο τα του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Η ΕΜΣΑ λοιπόν έλαβε 154 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ίδιο ποσό πήρε. Ο οργανισμός αρχικός είχε ζητήσει 198 εκατομμύρια λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό και άλλα στοιχεία. Και στη συνέχεια εξέτασαν τις δαπάνες, ε, ε, έλαβαν υπόψη και κάποιες αποταμιέσεις αποτελεσματικότερης χρήσης των κονδυλίων και με αυτό έκαναν μια αναθεωρημένη πρόταση. Η αναθεωρημένη πρόταση λοιπόν είναι 154 εκατομμύρια για τις παρούσες αρμοδιότητες για το επόμενο δημοσιονομικό ε, πλαίσιο, αλλά υπάρχει και το θέμα της επέκτασης των αρμοδιοτήτων για εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και εκεί το βλέπουν λίγο διαφορετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι για αυτές τις νέες αρμοδιότητες θα πρέπει να δοθούν 6 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ζητά 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο υπολογισμός του οργανισμού περιλαμβάνει παρακολούθηση, ε, διάθεση ε, στόλου και εγκαταστάσεις στον Αρκτικό και στα Κανάρια νησιά και σε κάποιες περιοχές της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ε, διεξάγει σωστά τα καθήκοντα που ζητήθηκαν από τον οργανισμό αυτό και με κατάλληλο τρόπο μάλιστα. Και όπως σας είπα, αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα δεν είναι κατά πόσον είναι καλό ή κακό, διότι είναι ήδη η λιμένη απόφαση και αποτελεί προτεραιότητά μας. Η σύστασή μου λοιπόν είναι να δοθούν 185,5 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον οργανισμό αυτό προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει και τη τα καθήκοντά του αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Έγινε μια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάσαμε και το ενδεχόμενο να υπάρχουν έσοδα από τον ίδιο τον οργανισμό ε, και την δυνατότητα να έχει κάποια εξοικονόμηση χρημάτων με την σωστή χρήση των σκαφών του. Και όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα αντικατοπτρίζονται και στις ε, τροπολογίες. Αν δεν κάνω λάθος η προθεσμία είναι 27 Ιουνίου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ε, θα σας ανακουφίζει αυτό κύριε Πρόεδρε γιατί νομίζω ότι αρκετά είπα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάνατε ένα λάθος. Ε, είπατε 185,5 εκατομμύρια λίρες. Εννοούσατε ευρώ έτσι δεν είναι. Ο κύριος Μπράντμπουρν και η κυρία Φώστερ θα καταχάρηκαν μάλλον, αλλά μάλλον εννοούσατε ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Τέιλορ για την έκθεσή του που είναι απόλυτα θετική. Είναι γεγονός ότι ο φορέας ναυτικής ασφάλειας έχει πάρει πολύ καλή υποστήριξη από την Επιτροπή μας και μια γενικά θετική στάση για τα καθήκοντά του και τις δραστηριότητες αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν οδηγεί την Κομισιόν να παρουσιάσει πάντα νέε αρμοδιότητες για ένα τέτοιο φορέα χωρίς τα μέσα να τα χρηματοδοτήσει τα νέα καθήκοντα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τους πόθους μας, με τις ελπίδες μας και με τις επιδιώξεις μας θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία και με το Συμβούλιο γιατί το Συμβούλιο πρέπει να καταβάλει και ένα τμήμα της χρηματοδότησης μέσω των δημοσιονομικών προοπτικών που εφέτος είναι οπωσφικές. Θέλω να κάνω μερικά πράγματα απόλυτα σαφή. Ο φορέας ασφάλειας στη θάλασσα από την αρχή γιατί έπαιξε κάποιο ρόλο στη δημιουργία του φορέα αυτού, είχε αποφασίσει με τη Γενική Συνένεση ότι δεν αρκεί να έχει κανείς ένα στόλο, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπήρχε και ένας στόλος, ένα κομμάτι του στόλου που ήταν διτής χρήσης, δηλαδή να λειτουργούν σε φυσιολογικές συνθήκες, αλλά επίσης να είναι έτοιμος αυτός ο στόλος να προστρέξει σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποια καταστροφή στη θάλασσα. Επομένως, όταν γίνεται ένα ατύχημα, ειδοποιείται ο φορέας ασφάλειας στη θάλασσα και ο φορέας θα πρέπει να κινητοποιήσει τα πλοία που βρίσκονται πιο κοντά στο ναυτικό αυτό ατύχημα και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα ρήπανσης κτλ. Αλλά κύριε Τέιλορ, αυτά δεν είναι δωρεάν. Εισπράττουν κάποιο αντίτιμο για αυτήν την ε, δραστηριότητα. Επειδή έχουν όλο και περισσότερα καθήκοντα, αυξάνει αυτό το κόστος λειτουργίας αυτών των ε, πλοίων και των υπηρεσιών τους. Και φυσικά πάντα οι υπηρεσίες τους είναι υπηρεσίες οι οποίες πληρώνονται. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα από ένα τρίτο γιατί δεν πρόκειται για έκκληση που γίνεται από ένα κράτος μέλος, αλλά όταν πρόκειται για μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί φυσικά γίνεται για λόγους αλληλεγγύης η βοήθεια προς κάποιο πλοίο τρίτης χώρας. Στο φυσιολογικό σύστημα πάντα ανακτά ο φορέας το κόστος αυτό. Γιατί το εμπλεκόμενο κράτος <coughs> για το λογαριασμό του οποίου γίνεται ο αγώνας κατά της πληρώνει το λογαριασμό. Αλλά η ανησυχία μας είναι ότι η διεύρυνση των καθηκόντων θα σημάνει και περαιτέρω κόστος. Γιατί στην περίπτωση ε, ενός πλοίου το οποίο πρέπει να ανασκευαστεί, θα πρέπει κάποιος να υπομειστεί το κόστος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα κάλυψης. Δεν μπορούμε να φέρουμε στα Κανάρια νησιά ένα αλλιευτικό πλοίο που είναι στον ε, γασκονικό κόλπο και να του ζητήσει κανείς να προστρέξει. Επομένως πρέπει να υπάρχουν κάποια πλοία τα οποία βρίσκονται κοντά σε τις περιοχές αυτές και τα οποία είναι σε επιφυλακή και επομένως για την επανασκευή τους χρειάζεται κάποιο κόστος να υπομειστεί η ΕΜΣΑ. Αλλά εδώ νομίζω πρέπει να έχουμε μια γενική συμφωνία. Ότι όταν υπάρχουν πάντα νέε αρμοδιότητε, και αυτέ οι νέε αρμοδιότητε είναι απαραίτητε λόγω των μεγάλων ατυχημάτων που είχαν γίνει στον, κόλπο, στον, συγγνώμη, στον κόλπο του Μεξικού που υπήρξε ένα ατύχημα σε μια πλατφόρμα εξόριξης ή μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα ε, στην ανοιχτή θάλασσα. Για όλες αυτές λοιπόν τις αρμοδιότητες θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες μεν προστασίας και παρέμβασης, αλλά να δούμε ποιο είναι το κόστος του στόλου που πρέπει να είναι σε επιφυλακή και ποιος είναι και ο τρόπος με τον οποίο εισπράττουμε το αντίστοιχο τίμημα για την παρέμβασή τους. Αυτό είναι λοιπόν το κλειδί του όλου εγχειρήματο. Σίγουρα θα βρεθούμε κύριε Τέλειο σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό με το Συμβούλιο και επομένως θα καταλάβετε ότι οι ικανότητε της ΕΜΣΑ θα παραμείνουν στο επίπεδο αυτού που θέλουν να πληρώσουν τα κράτη-μέλη και όχι παραπάνω. Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Τέιλορ για το έργο του, με το οποίο μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Στα χαρτιά η ΕΜΖΑ αποκομίζει νέες αρμοδιότητες. Πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου, αρμοδιότητες λοιπόν που τις δίνει το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Αλλά όπως ελέγχθηκε προηγουμένως δεν μπορούν να υπάρχουν νέες αρμοδιότητες χωρίς νέα χρηματοδότηση. Η ΕΜΣΑ είναι μια πραγματικά αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος υπηρεσίας. Δεν μπορούν να πούνε κάτι τέτοιο όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να μπορεί να έχει μια ε, πρόσβαση και μια παρέμβαση έγκαιρη για να αποτρέψει τη θαλάσσια ρήπανση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως όφελος υπερ, υπερ, ε, υπερβαίνει το κόστος το ετήσιο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν στην έμψη την απαραίτητη χρηματοδότηση για να φέρει σε πέρα σε αυτό το έργο. Η Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη καν τον ετήσιο πληθωρισμό, που δεν είναι βέβαια υπερβολικός, δεν είναι υψηλός αλλά μιλάμε εδώ για αυτά ε, σε εκατομμύρια τα οποία δεν υπολογίζονται σε αυτήν την περίπτωση. Η Κομισιόν είχε πάρει 154 εκατομμύρια στην τελευταία περίοδο και τώρα παίρνει 6 εκατομμύρια παραπάνω για την επόμενη επταετή περίοδο. Αυτό δεν είναι σωστό γιατί όπως σας είπα είναι τα 7 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Γι' αυτό συμφωνώ με τη θέση του, ε, του εισηγητή για το ποσό αυτό των 158 εκατομμύριων. Το ερώτημα είναι και τι σκοπούς θα εξυπηρετήσει αυτό το χρήμα. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διεύρυνση των, δια... των αρμοδιοτήτων γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μονάχα στις ε, ίδιες τις πλατφόρμες και όχι στην ευρύτερη περιοχή του αρμοδιότητα. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμός γιατί δεν μπορεί κανείς να πάει σε μια πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσει τα παραδοσιακά ε, μέσα αντιμετώπισης των ε, ρηπάνσεων. Θα πρέπει να μισθωθούν νέα πλοία. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει και μία προσθήκη προσωπικού και τεχνογνωσίας και κατάρτισης του προσωπικού. Εμείς υπολογίζουμε ότι χρειάζονται 98 δισεκατομμύρια, ε, η ΕΜΣΑ θέλει 198, ίσως μπορούμε να βρούμε κάπου μια συμβιβαστική λύση σε αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα είναι σημαντικό. Όπως λέμε, αυτός ο οποίος ζητάει κάτι το πληρώνει κιόλας. Εδώ δεν πρόκειται για τον ε, κύριο Κάλλας και τις υπηρεσίες του, πρόκειται για τον Επίτροπο Έτεγκερ, ο οποίος πρέπει να φέρει τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί λοιπόν οι αρμόδιες ε, υπηρεσίες για τα ενεργειακά θέματα δεν θα πρέπει να συμβάλλουν και ο προπολογισμό για την ενεργειακά δεν θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε Μπιλμπάου. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τέιλορ για την προσπάθειά του και εγώ θα είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα επιχειρήματα ούτως ή άλλως τα είπαν οι συνάδελφοι, ο καθένας με τον τρόπο του φυσικά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια αλλαγή στον οργανισμό, του ανατέθηκαν νέα καθήκοντα και τα νέα καθήκοντα όπως βλέπουμε και μας λένε και τα στοιχεία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτός και αν αυξηθεί ο προπολογισμό. Πρέπει να πω ότι η ιστορία του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και η δημιουργία τους έχει προκύψει από μια κρίση, διότι οι καταβολές του οργανισμού είναι από το Έρικα, το ναυάγιο του Πρεστής ε, και τα όσα συνέβησαν στον κόλπο του Μεξικού. Σιγά σιγά λοιπόν τροποποιούμε και βλέπουμε πόσο ανάγκη έχει αυτός ο οργανισμός και αυξάνουμε τα καθήκοντά του όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να ε, διορθώσουμε. Τροποποιώντας λοιπόν τα καθήκοντα του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα πρέπει να υπάρχει και αύξηση αντίστοιχα στον προπολογισμό. Και να απαντήσω και στον εισηγητή και να του πω ότι δεδομένου των δυσκολιών που έχουμε με τον ε, προπολογισμό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πούμε στο Συμβούλιο ότι αυτοί ενέκριναν τι νέε αρμοδιότητε και δεν μπορεί να διεξάγει τα καθήκοντά του οργανισμό επιπλέον κονδύλια. Και στην προηγούμενη έκθεση είχαμε ήδη συμπεριλάβει και τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη ανάλυση των τεχνικών στοιχείων, τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές ε, και την καινοτομία προκειμένου ε, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών και να εφαρμόζονται οι πρακτικές για να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις της ε, θαλάσσιας ρήπανσης. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς και μόνο για αύξηση του προσωπικού. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση, τις βέλτιστες πρακτικές και την συνεχή επιμόρφωση του προ προσωπικού που ε, εργάζεται στον οργανισμό. Και το θέμα είναι τι θα γίνει αν υπάρξει μια νέα καταστροφή η οποία πάλι θα μας ε, καταλάβει εξαπίνης. Ε, τι θα γίνει, ποιος θα είναι υπόλογος επειδή δεν συμπεριλέβανε στον προϋπολογισμό επιπλέον κονδύλια για να διεξάγει τα καθήκοντά του. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την άγουσα του εισηγητή. Θα παρουσιάσουμε και εμείς κάποιες τροπολογία με στόχο να βελτιωθεί το θέμα της κατάρτισης, τη βελτίωση των δεδομένων, οι καλές πρακτικές, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και προς αυτό το σκοπό ελπίζω ότι όπως είπαμε και στην προηγούμενη έκθεση θα καταλήξουμε σε μια ε, συνενετική απόφαση. Ευχαριστώ κύριος Μπράτπορν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους, όπως μας είπε και ο κύριος Τέιλερ, ότι αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο το εάν και κατά πόσο θα αναλάβει νέε αρμοδιότητε ο ε, Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Αυτό έχει συμβεί. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση. Θα περιοριστώ λοιπόν στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Από ό,τι φαίνεται θα σταθώ μόνος ε, εδώ γιατί διαφωνώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί νέα χρηματοδότηση. Εφόσον, όπως όλοι γνωρίζουμε, στις διαπραγματεύσεις για το πολιτισμο νομικό πλαίσιο, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει περικοπή του προπολογισμού και εδώ εμείς ζητούμε και άλλα χρήματα για έναν οργανισμό. Όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι και ε, μεγάλος αυτών των οργανισμών, αλλά, αλλά στα θέσω σε μια βάση. Όταν εξετάζουμε αυτούς τους προπολογισμούς ε, βλέπουμε ότι αυτομάτως ναι πρέπει να γίνει αύξηση εδώ, αύξηση εκεί. Ε, είναι μια ληστητική αντίδραση. Δεν κοιτάζουμε άλλες ε, επιλογές όπως θα μπορούσαμε ας πούμε, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε σε άλλους τομείς, σε άλλους τομείς του προπολογισμού όπως ανέφερε και ο Σοσιαλδημοκράτης συνάδελφος. Εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και συνέχεια βλέπω ε, ποσά που δεν απορροφώνται. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζουμε ευρύτερα αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια από άλλους προπολογισμού, αν μπορεί να γίνει μετάβαση, μεταφορά κονδυλίων από, τον ένα, από το ένα τμήμα στο άλλο, πριν περάσουμε στη διαδικασία όπου ζητάμε περισσότερα κονδύλια. Αυτό θα ήθελα να δω και το είδα σε αυτήν την έκθεση. Πριν από καιρό, έβλεπα τη συνεργασία με τις ε, τοπικές αρχές. Εκεί ε, περισσότερες αρμοδιότητες, δεν ζητούσαμε κάθε φορά παραπάνω χρηματοδότηση, εξοικονομούσαμε πόρους από άλλα τμήματα. Και αυτό θα ήθελα να συμβεί εδώ. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα θέσπιση μηχανισμών όπου και ο ίδιο ε, ο οργανισμό ε, μπορεί να συλλέγει ε, πόρου από τρίτου φορεί. Όμω αυτό θα πρέπει και πάλι να συμπεριληφθεί στον ευρύτερο προπολογισμό. Γιατί τα χρήματα που έχουμε στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πάσα πιθανότητα θα μειωθούν, θα συρρυκνωθεί ο προπολογισμό και έτσι θα πρέπει και εμεί να είμαστε ρεαλιστέ έτσι, δυστυχώ κύριε Τέλορ, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη σύστασή σα. Εγώ θα ήθελα μάλιστα μείωση ε, των προπολογισμών τέτοιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένη και στη ΣΕΜΣΑ. Ο κύριος Ζήκη, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Γιατί ο προλαλής ε, ανέφερε αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Γιατί έχω μια ελαφρώς διαφορετική θέση. Ε, ως εισηγητής για τον προπολογισμό του 2014 ήθελα μόνο να πω ότι κατανοώ τα επιχειρήματα του εισηγητή και της ε, πλειονότητας των σκιωδών. Συμφωνώ βέβαια με τα όσα υπόθηκαν, αλλά αντιθέτως με τον προλαλήσαντα εγώ είμαι υπέρ αυτών των οργανισμών, όμως ε, πράγματι αυτά χρηματοδοτικά τους μέσα θα πρέπει να θα μειωθούν στη γραμμή 06 των μεταφορών και για να δώσουμε περισσότερα χρήματα στον οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από αλλού. Και υπάρχουν και, άλλες, και άλλοι οργανισμοί που θα αναλάβουν περαιτέρω αρμοδιότητες όπως ε, για τους υδροδρόμου. Και υπάρχουν και άλλες δημοσιονομικές εξελίξεις. Συμφωνώ πλήρως επί τη βάση με τον εισηγητή, όμως υπάρχει ένα ζήτημα βάσης προπολογισμού, κάτι το οποίο δεν έχει επιληθεί ακόμα και θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Κύριε Φλάκενστάιν, ζητάτε εντόνως το λόγο, να είστε σύντομος παρακαλώ. Τρεις φράσεις. Εμείς έχουμε ήδη αποφασίσει γιατί θέλουμε να εμποδίσουμε να, κοστίσει, να το κάνει αυτό η έμψη γιατί αλλιώς θα κόστιζε περισσότερο. Δεύτερον, αν θέλετε να το κάνει αυτό η ΕΜΣΑ, να μας πείτε από πού θα εξοικονομήσουμε τα χρήματα, από ποιο άλλο φορέα, αλλά δεν μπορεί να αναλαμβάνει κοντά χωρίς χρηματοδότηση. Και τρίτον, αν είναι τα πράγματα όπως λέτε κύριε Ερικέ, πρέπει να πούμε στους ε, πολίτες, κάναμε λάθος, θέλαμε να κάνουμε όλες αυτές τις περαιτέρω ενέργειες με την έμψα, αλλά δεν θα δώσουμε λεφτά ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για τον εξοπλισμό για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι αρμοδιότητες. Κυρία Μπέρκ από την Κομισιόν. Σύντομα μπορείτε κυρία Μπέρκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τέιλο και όλα τα μέλη για τις συζητήσεις που είχαμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι ότι αυτή είναι μια πρόταση του προϋπολογισμού και το θέμα δεν είναι το ορθό ή το λανθασμένο της πρότασης. Η ΕΜΣΑ κάνει σωστά την εργασία του. Φυσικά η Κομισιόν αντιμετωπίζει δυσκολίες με το να παρουσιάσει αυτή την πρόταση, γιατί φυσικά καταγράψαμε αυτά τα οποία ζητά ο νέος κανονισμός για την ΕΜΣΑ, αλλά είναι φανερό ότι αυτοί οι νέοι, οι νέες αρμοδιότητες για την ΕΜΣΑ δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις ε, διαπραγματεύσεις, δεν πρέπει να επηρεαστούν μάλλον με τις διαπραγματεύσεις για τις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν στον εαυτό μας είναι ότι συνολικά ο προϋπολογισμός για τους αποκεντρωμένους φορείς θα μείνει σταθερό στα επόμενα 7 χρόνια. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι η βάση της πρότασής μας, και έτσι εξασφαλίζουμε ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών του φορέα αυτού της ΣΕΜΣΑ και αν δεν θέλουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες εφόσον εσείς, εσείς δεν θέλετε να θέσουμε σε δυσκολία τους άλλους λειτουργικούς φορείς τότε πρέπει να παγώσουμε και τα λειτουργικά κονδύλια, ε, κονδύλια για την απορρίπανση που μας φέρνει στα 154 εκατομμύρια τα οποία έχουμε αναφέρει. Βέβαια η έμψα παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά όλο περισσότερο, καταφέρει να έχει συμβόλαια τα οποία είναι φθηνότερα, να αποκομίζει καλύτερες συνθήκες και να είναι πιο αποτελεσματική με, την, με τα χρήματα που έχει στη διάθεσή Αυτό πρέπει να μπει στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικές και με τη σταθεροποίηση του προπολογισμού έχουμε απλώς κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε, να κάνουμε ένα facing in αυτών των νέων δραστηριοτήτων και είπαμε για αυτά τα λίγα λεπτά δεν είναι δυνατό να μπούμε και στην ε, ε, να έχουμε και νέα πλοία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ε, για τους στόχους αυτούς, οπότε είπαμε η ΕΜΣΑ τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει τις διαλυτικές ουσίες που είναι η τελευταία καταφυγή αν έχετε μεγάλες κοιλίδες ρήπανσης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αλλιώς. Με την πρόταση αυτή λοιπόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ως αρχές του προϋπολογισμού γιατί περί αυτού πρόκειται. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά θέματα μαζί με την ΕΜΣΑ. Εάν κάποια από τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν τέτοια προβλήματα και θέλουν πληροφορίε για να καταθέσουν τροπολογίες, αλλά αυτή τη στιγμή για τις 11 τροπολογίες που έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί, εγώ, εγώ έχω εξηγήσει γιατί καταλήξαμε με ένα περιοριστικό προϋπολογισμό. Όλα τα άλλα βέβαια μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε θετικά. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια αναδιατύπωση για ορισμένα πράγματα, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Συμβουλίου σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα κύριε Τέιλορ πριν πω τις προθεσμίες. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Άκουσα τι είπε ο κύριος Μπράτμπουρν. Το να λάβουμε κονδύλια από άλλες γραμμές προϋπολογισμού και να αυξήσουμε αυτόν τον προπολογισμό δεν είναι πράγματα τα οποία αποκλείουν το ένα το άλλο. Πάντα υπάρχει τρόπος. Έχω εργαστεί και εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση για πάρα πολλά χρόνια και ε, γνωρίζω πώς να εξετάζω τον προπολογισμό με πιο δημιουργικό τρόπο. Υπάρχουν ε, πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλη τα οποία προέρχονται από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αν δείτε τις συστάσεις μου θέλουμε απλώς επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια. 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν δείτε την κοστολόγηση για τα μέτρα απορρίπανσης, το κόστος μόνο και μόνο για τους δορυφόρους είναι 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αντισταθμιστούν, αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε λίγο πιο δημιουργικά τα επιχειρήματά μας και πρέπει να είμαστε και λίγο πιο εφευρητικοί να δούμε πού μπορούμε να βρούμε κονδύλια. Απλώ βλέπω στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 27 Ιουνίου. Ψηφοφορία 17 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για την Ολομέλεια. 27 Ιουνίου, 17 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, η μήνυα ακρόαση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αν δεν κάνω λάθος, όλοι εδώ είμαστε. Να ξεκινήσω λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ακόμα εν ανεμονή της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συστάσεις ε, του ε, οργανισμού για την, τον Ευρωπαϊκό Ουρανό και ξέρετε ότι ήμουν και εγώ εισηγητής στη σχετική έκθεση και θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτή η πρόταση είναι βάση επιτροπολογίας επομένως δεν μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Ε, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τις συστάσεις της, είτε θα ε, εγκρίνουμε είτε θα απορρίψουμε την πρόταση. Και αν καταψηφίσουμε την πρόταση, τότε το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή οι υφιστάμενοι περιορισμοί στις πτήσεις, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Αυτό και να είναι απόλυτα σαφής, διότι νομίζω ότι υπήρξε μια παρανόηση για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Να υπενθυμίσω επίσης ε, στους συναδέλφους ότι αυτή είναι μια έκθεση η οποία δεν γίνεται για διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ε, και τις συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι θέμα των κοινωνικών εταίρων που ασχολούνται με το θέμα. τι θα κάνουμε. 10 λεπτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 λεπτά για τις αεροπορικές εταιρείες, ε, δηλαδή ε, από 5 λεπτά ο καθένας. Ε, μετά θα δώσουμε 5 λεπτά για τις εθνικές αρχές, 5 λεπτά για τους εμπειρογνώμονες για τη διαχείριση και 5 λεπτά για την σας στο τέλος και μετά θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωταποκρίσεων από πλευράς ε, συναδέλφων. Επίσης να σας πω ότι δέχθηκα πάρα πολλά αιτήματα για να μιλήσουν ε, διάφοροι στη συγκεκριμένη ακρόαση. Αν δεχόμουν ε, να μιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν, μέχρι τον Ιούλιο θα κάναμε ακρόαση για το συγκεκριμένο γεγονός. Επομένως πρέπει να επιλέξω κάποιους. Εάν κάποιοι ενοχλούνται λυπάμαι πολύ αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ξεκινώντας λοιπόν... Να δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση MOVE, τον κύριο Μπόλτιν, ο οποίος είναι Διευθυντής ε, Αεροπλοείας και Διεθνών ε, Μεταφορών. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα φροντίσω να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα, διότι πρωτίστως θέλω να ακούσω τι έχουν να πούνε οι υπόλοιποι σε αυτή τη τόσο σημαντική ακρόαση. Σα ευχαριστώ που τη διοργανώσετε και σα ευχαριστώ που προσκαλέσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι γίνεται αυτή η ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών, διότι εδώ είναι το θέατρο των επιχειρήσεων στο οποίο συζητούνται όλα αυτά τα θέματα και έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν και ε, προφανώς είναι πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω λίγο την κατάσταση. Πού έχουμε φτάσει στη διαδικασία της πρότασης των αλλαγών στον ε, παρόν καθεστώς ε, περιορισμού στις πτήσεις και να σας πω ότι κυρίως μας ενδιαφέρουν τρία πράγματα. Ασφάλεια, ασφάλεια και πάλι ασφάλεια. Δεν μας ενδιαφέρουν ε, οι συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες για τους κυβερνήτες των αεροσκαφών και το προσωπικό τους αεροσυνοδούς. Μας ενδιαφέρουν και αυτά, αλλά δεν μας αφορούν εδώ. Ούτε μας ενδιαφέρει το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες που είναι εξίσου σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο αυτής της νομοθεσίας. Και νομίζω ότι δικαίω λέω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα τουλάχιστον και εμείς και οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες μας βρίσκει σύμφωνους. Όλοι θεωρούμε το πιο σημαντικό την ασφάλεια. Και ο στόχος της ασφάλειας θεωρούμε ότι καλύφθηκε από τις προτάσεις που έγιναν στη γνωμοδότηση της ΕΑΤΑ ΕΑΣΑ τον Οκτώβριο του 2012 μετά από τρία χρόνια διαβουλεύσεων με διαφόρους ενδιαφερομένους και χαίρομαι που είναι εδώ και ε, κάποιοι εξ αυτών και θα μιλήσουν αργότερα. Ε, όταν συζητήθηκαν στην Αρμόδια Επιτροπή έλαβαν και ε, ε, σχετικά θετική ανταπόκριση, αλλά πρέπει να απαντηθούν και κάποια ερωτήματα. Υπήρχε εξαιρετική συνεργασία με τους ενδιαφερομένους για να γίνουν προτάσεις οι οποίες πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρές. Μα ενδιαφέρουν διάφορα πράγματα τα οποία εξέφρασαν κυρίω οι συνδικαλιστικοί φορεί για αρκετά ζητήματα. Για τα ε, καθήκοντα του αεροδρομίου, το ε, ε, προσωπικό ασφαλείας, ε, τις κατάλληλες εκθέσεις και νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στον τομέα αυτό. Και έχει γίνει και κάποια πρόοδος, θεωρώ, και έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις Μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τους χρόνους αναμονής εκτός χώρου αεροδρομίου, τι γίνεται με τους ε, διαφόρους χρόνους ε, των πληρωμάτων και έχουμε συζητήσει το θέμα αναλυτικά με τις αεροπορικές εταιρείες και έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα για την ασφάλεια και αν δεν κάνω λάθος ε, θα ακούσουμε την άποψη και των ΜΕΝ και των ΔΕ για τις ανησυχίες που έχουν για το θέμα αυτό. Δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο της επίσημης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι στα σκαριά όμως και σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε στην Ρυθμιστική Επιτροπή της ΕΑΣΑ στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε να λάβουμε και τη θετική τους γνώμη στις 11 Ιουλίου. Κατόπιν, αυτή τη στιγμή συγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν ε, τρει μήνε βάση του συστήματο για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την πρόταση, το οποίο χοντρικά σημαίνει ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο, ε, στο οποίο συμφωνούν κατά την άποψή μου οι περισσότεροι, ότι ήγηκε πλέον η ώρα, κύριε Πρόεδρε, να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Είναι ελάχιστα τα θέματα τα οποία έχουν μελετηθεί τόσο επισταμένα και έχουν ε, ληφθεί αποφάσεις από αυτόν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ζητά κανεί συγγνώμη διότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και παθιάζει τον κόσμο. Θεωρούμε λοιπόν πλέον ότι έχουμε μία εύρωστη πρόταση που θα κάνει ακόμα πιο ασφαλή τις πτήσει στην Ευρώπη και εγώ είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πιο προστατευτικά μέτρα γιατί είναι πιο αυστηρά από τα μέτρα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι θα αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο τη ε, ασφάλεια και τη προστασία στα περισσότερα κράτη-μέλη. Κάποια άλλα θεωρούμε ότι θα δώσουν το επίπεδο ασφάλεια το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό που παρέχουν κάποια κράτη-μέλη και παρεπιπτόντω και αντίστοιχο των ΗΠΑ. Δεν είναι πανομοιότυπο, διότι αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο εμεί και οι Αμερικανοί, αλλά θεωρούμε ότι το θέμα τη ασφάλεια μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ένα συνδυασμό ε, συγκεκριμένων μέτρων. Η έκκλησή μου λοιπόν σήμερα είναι να μην καθυστερήσουμε καθόλου περισσότερο το θέματα αυτά. Πρέπει να εγκριθούν αυτά τα μέτρα και να εφαρμοστούν, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι προ όφελο των ε, πολιτών μα, των επιβατών και των πληρωμάτων. Πριν ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, ε, να σας πω ότι ε, εφαρμόστηκαν ε, πολλά επιστημονικά στοιχεία. Η ΆΣΑ τα χρησιμοποίησε πλήρως όταν παρουσίασε τη γνωμοδότησή της και πιστεύουμε βαθύτατα ότι κάνουμε προτάσεις οι οποίες σέβονται απόλυτα τις επιστημονικές ενδείξεις. Να σας επιστήσω όμως την προσοχή στο εξή. Κάποιες από τις μελέτες οι οποίες γίνονται και αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι είναι πολύτιμες για να κατανοήσουμε σημαντικά στοιχεία του συστήματος περιορισμού των πτήσεων, ε, μπορεί να παρανοηθούν εάν τα συζητήσουμε εκτός πλαισίου. Καλό λοιπόν θα ήταν να γνωρίσουμε ότι αυτές τις εκθέσεις δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε ως βάση για να αξιολογήσουμε τη συνολική αποτελεσματικότητα του ε, αμαλγάματος αυτού των μέτρων που προτείνουμε. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει μια πλήρης εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος και αυτό προτάθηκε και στην αρχική γνωμοδότηση της ΕΑΣΑ. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι για πρώτη φορά δεν έχω υπερβεί και το χρόνο μου, ε, προσβλέπω στη συζήτηση, ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω και σύντομα στο τέλος και όπως σας είπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ για να τίνει ευήκονους. Πρωτού περάσω στις απόψεις των αεροπορικών εταιριών, θέλω να χαιρετήσω την ομάδα που έχει προσκαλέσει ο κύριος Κράμερ από, την, ε, από το Βερολίνο και το Βραδεμβούργιο. Καλώς ήλθατε λοιπόν εδώ. Ελπίζω ότι θα χαρείτε την επίσκεψη σας εδώ στους Βρυξέλλες. Δίνω τώρα το λόγο στις αεροπορικές εταιρείες και ξεκινώ με τον κύριο Βίνσεν Ντεμπρόι, ο οποίος είναι ο Γενικός ε, Διευθυντής της Ένωσης των Αεροπορικών Φορέων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι μας καλέσατε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας στην τόσο σημαντική σας εταιρεία. Το να είναι να μην είναι σε κατάσταση υπερβολικής κόπωσης το πλήρωμα καμπίνας και το πλήρωμα του πιλωτηρίου είναι ε, πολύ σημαντικό. Αν νομίζετε ότι είναι ακριβές αυτές οι υπηρεσίες, τα πληρώματα, τότε δοκιμάστε με ατυχήματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια κοινή ευθύνη των αεροπορικών εταιριών και των πληρωμάτων. Οι αεροπορικές εταιρείε πρέπει να ακολουθήσουν ε, αυστηρούς κανόνες και τα μέλη του πληρώματος έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν σωστά τις απαιτήσει ανάπαυσης και να μην είναι κουρασμένοι όταν έρχονται για να συνεχίσουν τις βάρδιες τους. Η πρόταση λοιπόν αυτή για τον χρόνο πτήσης είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαβούλευσης με, τους, ε, με τα εργατικά συνδικάτα και τις εθνικές αρχές η άποψη της ΙΑΚΑ βασίζεται σε περίπου 50 επιστημονικές μελέτες και τους εθνικούς κανόνες και τις λειτουργικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Επί τη βάση αυτής της πρότασης η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα για χρόνο πτήσης, πιο αυστηρά και από την ε, αμερικανική ρύθμιση και από τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα σε κάποιες χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία κτλ και πρέπει να τονίσω ότι και οι προηγούμενοι κανόνες εξασφάλιζαν την ασφάλεια. Η πρόταση αυτή επίσης είναι αντίστοιχη με τους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου και πάντα θεωρούν οι εμπλεκόμενοι ότι είναι ένα είδος σημείο αναφοράς το Ηνωμένο Βασίλειο και οι αρχές ε, πολιτικής αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν χαιρετήσει αυτές τις προτάσεις. Τέλος, η πρόταση της ΙΑΚΑ είναι πιο αυστηρή και από τους κανόνες της Αμερικανικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Αεροπορίας. Δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια δώσανε συγκινησιακό χαρακτήρα σε αυτή την συζήτηση και έχουν παραπληροφορήσει για τα θέματα αυτά έχουν αποφασίσει να διαλέξουν επιλεκτικά αυτά τα οποία τους βολεύουν για ορισμένα θέματα και πολλές φορές αναφέρουν επιστημονικές και ψευδοεπιστημονικές εμπειρογνωμοσύνης εκτός πλαισίου για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Είναι πολύπλοκα τα θέματα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, πάντα πρέπει να τις βλέπουμε όμως αυτές ως ένα πακέτο. Η ασφάλεια δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με το να απλοποιήσουμε ένα πολύπλοκο θέμα και να καλλιεργήσουμε μια ατμόσφαιρα φόβου οι αρμόδιοι για τους κανόνες ασφάλειας είναι υποχρεωμένοι να θεσπίσουν κανόνες για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, αλλά όχι να ρυθμίσουν κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες. Εξάλλου και γι' αυτό το λόγο εσείς είσαστε αρμόδιοι για το θέμα αυτό και όχι η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνθήκες εργασίας των πιλότων και του πληρώματος είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ εταιριών και εργατικών συνδικάτων επί τη βάση της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μας αυτή δεν το τροποποιεί αυτό. Οι συνθήκες εργασίας όμως των αεροπορικών εταιριών θα πρέπει να συμμορφώνται με τα πιο αυστηρά όρια τα οποία θεσπίζονται από την πρόταση της Κομισιόν. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ ισορροπημένη, δημιουργεί κάποιο πρόσθετο κόστος για μεγάλες εταιρείες, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι λόγος για να το θέσουμε ένα αμφιβόλο αυτό το νέο καθεστώς από 11 ώρες 45 λεπτά που ισχύουν τώρα έχει μειωθεί το όριο εργασίας ε, σε 11 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι πτήσεις που ε, ξεπερνούν τις 9 ώρες χρειάζονται ένα τρίτο πιλότο. Οι ε, ορισμένοι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι αυτό δεν φτάνει και θέλουν να θέσουν το όνομα σε 10 ώρες. Αλλά αυτές είναι απόψεις οι οποίες δεν ε, εδρεώνονται σε επιστημονικές θέσεις για την ασφάλεια. Επίσης έχουν υπάρξει λανθασμένες ε, πληροφορίες γιατί θεωρούν οι ερωσμένοι μπλεκόμενοι γιατί θεωρούν το πλήρωμα δεν μπορεί να κοιμάται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό είναι μια τελείως θεωρητική αντιμετώπιση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θεωρεί ότι όταν κάποιος είναι σε επιφυλακή δεν είναι σε θέση να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί. Και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Το ίδιο πράγμα γίνεται όταν είναι κανείς επιφυλακή στο σπίτι του. Είναι πάντα έτοιμος να έρθει στην εργασία του ακόμα και εάν ε, ξεκουράζεται. Θέλω να κλείσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι οι νέοι αυτοί κανόνες θεσπίζουν ένα καθεστώς το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή αεροπορία και θα είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων επιβατών γιατί όλες οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Είναι καιρός λοιπόν να δεχτούμε αυτούς τους ε, κανόνες και να μην επηρεαστούμε από ένα κλίμα φόβου που δημιουργείται από ορισμένου και από την παραπληροφόρηση που δημιουργούν. Next, Mr. Eric Director of Safety Ευχαριστούμε. Επόμενο ο κύριο από τη Διεθνή Ένωση για τι Ναυλωμένε Πτήσει. Παρακαλώ για πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, εξωτήμα μέλη τη Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού, σα ευχαριστούμε που προσκαλέσατε την Ένωσή μα για τους νέους κανόνες. Εγώ σα μιλώ και ως πρόεδρος ε, ε, του συμβουλευτικού οργάνου για τα πρότυπα της ε, ΙΑΚΑ. Τον συγγνώμη. Βεβαίως ε, και συμμετέχουμε σε όλες τις εργασίες. Γι' αυτό ακριβώς ε, οι αερομεταφορείς της Ένωσής μας είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τους νέους αερομονισμένους κανόνες. Εφόσον η πλειονότητα των, Ευρωπαίων καταναλωτών κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, το κόστος είναι διπλάσιο σχέση με το χειμώνα. Ενώ τα πρότυπα προσπαθούν υποτίθεται να κατανείμουν ισόποσα σε όλο το χρόνο το κόστος, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε ε, μηνιαία βάση. Για να γίνει αυτό, το άκα πρέπει να κάνει εκπεριτροπής ε, διεργασίες ε, αρκετές φορές την ημέρα. Ε, και ακολουθείται η κόκκινη γραμμή σε σχέση με την μπλε γραμμή που αφορά τις ευρωπαϊκές γραμμές. Η ΆΚΑ μεταφέρει τους ευρωπαίους καταναλωτές οπουδήποτε θέλουν για τις καλοκαίρινες διακοπές. Επομένως καλύπτουμε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς. Πολλοί προορισμοί καλύπτονται μόνο μία-δύο φορές την εβδομάδα. Ε, με οικονομική θέση μάλιστα. όμως με τα νέα πρότυπα θέλουμε περισσότερες ε, πτήσεις και αυτό δημιουργεί προβλήματα και για τους ε, καταναλωτές αλλά και για τα πληρώματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη καν τον οικονομικό αντίκτυπο για τον εμπορευόμενο. Η ΆΚΑ μπορεί να μεταφέρει τους ευρωπαίους καταναλωτές προς τους, ε, προς προορισμούς διακοπών τους και στην τιμή που μπορούν να, πληρώσουν. Ε, οι θέσεις business δεν είναι κατάλληλες για, το, για, για τον τομέα των διακοπών οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να γίνουν οικονομικά βιώσιμοι μόνο αν έχουν πλήρες κρατήσεις ή σχεδόν πλήρες κρατήσεις. Παρά τις, ε, την εξαιρετική εργασία εδώ και δεκαετίες, τα προτινόμενα πρότυπα θα εμποδίσουν ε, τη συνέχιση των ε, κτήσεων με οικονομικές θέσεις. Η ΆΚΑ χαιρετίζει το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για τις ε, εγκαταστάσεις ανάπαυσης εντός του αεροσκάφους δεν συμπεριλαμβάνονται στους ίδιους εφαρμοστικούς κανόνες ε, γιατί απαιτούνται ε, περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία. Το 60% όλων των πτήσεων της ΕΑΚΑ τη νύχτα υπερβαίνουν τις 10 ώρες και δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν υπήρχε και ένα επιπλέον όριο όπως προτείνεται στους νέους κανόνες FDL να σημειώσουμε ότι αυτές οι πτήσεις πραγματοποιούνται από τα narrow body aircraft και δεν μπορούν να αυξηθούν λόγω της έλλειψης χώρου μες στο αεροσκάφος. Αν υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί θα έχουμε τεράστια, τεράστιες ζημίες για ορισμένε από τις εταιρείες μας. Κάποιες από αυτές θα πληγούν κατά 100% οποιοδήποτε επιπρόσθετο όριο δεν μπορεί να αναλυφθεί από άλλον εμπορευόμενο για τους λόγους που σας ανέφερα. Έτσι θα υπάρξουν ζημίες για όλους. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Εμείς καλούμε την Επιτροπή σας να εξετάσει σοβαρά ε, τον αντίκτυπο των προτινόμενων κανόνων που θα έχουν στον θεριστικό ε, ε, τομέα σε περιοχές όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, αν δεν υπάρχουν πλέον πτήσεις προς αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να υπάρξουν έντονες διαβουλεύσεις και με την ΙΑΚΑ και με διεθνείς άλλους οργανισμούς. Ως πρόεδρος ε, της, ε, του γνωμοδοτικού οργάνου για την ΕΑΣΑ μπορώ να ε, χαιρετήσω τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης, όμως θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να προσαρμοστούμε στα νέα πρότυπα. Χαιρετίζουμε παρόλα αυτά την πρόταση για την αξιοπιστία την, της ΕΑΣΑ. Εμείς λοιπόν θέλουμε οι τελικοί κανόνες να είναι ταυτόσιμοι με τη γνωμοδότηση της ΕΑΣΑ. Ελπίζουμε η Επιτροπή σας να εξετάσει με προσοχή ε, τον επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και ε, στις αερομεταφορές αλλά και στον τουριστικό τομέα οποιασδήποτε τροποποίησης που προτείνετε πριν αναλάβετε και υιοθετήσετε απόφαση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους των συνδικάτων, καταρχάς η κυρία Ελισαμπέτα Τσίκα από το ETF. Παρακαλώ, έχετε πέντε λεπτά. Κίκα. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Να ευχαριστήσω τον Brian Simpson, πρόεδρο της Επιτροπής που κάλεσε την ETS ε για να μιλήσει για τους περιορισμούς της πτήσης. Λέγομαι Ελιζαμπέτα Κίκα, είμαι μέλος της Αλιτάλια εδώ και 26 χρόνια και είμαι και επικεφαλής του πληρώματος καμπίνας του ETF ε και προσωπούμε ε, πάρα πολλές οργανώσεις ε, πανευρωπαϊκά. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα επισέλθω κατευθείαν στο προκείμενο. Καταρχάς ε, βελτιώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν βελτιώσεις στον τελικό κανονισμό όπως μας υποσχέθηκε. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει όλες αυτές τις βελτιώσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν στην καλύτερη ασφάλεια του αεροπλάνου. Ε, χρόνος αναμονής ε, για το πλήρωμα, να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, να υπάρχουν ε, επιφυλακή στο αεροδρόμιο, νυχτερινές πτήσεις, κατάλληλη διαχείριση, οδηγία για το χρόνο εργασίας, να μην υπάρχει ρήτρα υπαναχώρησης και να υπάρχει και ρήτρα αναθεώρησης. Τώρα, για το πλήρωμα καμπίνας και για τους κυβερνήτες είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Αν οι βελτιώσεις αυτές δεν συμπεριληφθούν στην κανονισμό θα δημιουργηθεί κούραση και αυτό θα είναι εις βάρος της ένα από τα βασικά στοιχεία της οργάνωσής μας είναι ο χρόνος ε, επιφυλακής. Εδώ κατανοούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον κανονισμό αυτό το πλήρωμα θα βρίσκεται σε επιφυλακή μέχρι και 16 ώρες και μετά θα φεύγει για κάποια πτήση για το μέγιστο αριθμό των επιτρεπόμενων ωρών. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ε, χωρίς ύπνο για 16 ώρες και μετά θα εργαστούν. Αυτό είναι ασφάλεια και θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το μέγιστο δυνατό χρόνο και να το συνδυάσουν με το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο επιφυλακής και αυτό γίνεται μόνο για οικονομικούς λόγους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε την ασφάλεια ούτε τις επιστημονικές ενδείξεις. Δεν εμφανίζεται ε, κάποιο ανώτατο όριο στον κανονισμό και οι 16 ώρες ε, ε, είναι λένε το ίδιο όρο που εφαρμόζεται με τη ΣΥΠΑ ο χρόνος επιφυλακής ε, δεν ε, προσμετράται στη μείωση του χρόνου πτήσης και αυτό φυσικά είναι εις βάρος της κούρασης ε, του πληρώματος. Υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούν τώρα οι Ευρωπαίοι αερομετεφερείς ε, κάποιες πτυχές που αφορούν κυρίως την εξοικονόμηση χρημάτων και να μην λαμβάνουν υπόψη την κούραση. Τα προβλήματα που προκύπτουν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι οι κερδοσκόποι ε, των αεροπορικών εταιριών θα προσπαθήσουν να εργάζονται στις παρυφές της νομιμότητας και νομίζω ότι το πλήρωμα δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς ύπνο και να είναι μετά σε κατάσταση να εργάζεται. Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να μείνει ξύπνιος για 16 ώρες και θα πρέπει μετά να κοιμάται 8 ώρες. Αλλιώς αποδεικνύεται από τις υποστημινικές ενδείξεις ότι ε, η κρίση του καθενός επηρεάζεται πάρα πολύ αν έχει μείνει 16 ώρες χωρίς ύπνο. Και τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να ισχύουν λοιπόν και για το χρόνο επιφυλακής και στο αεροδρόμιο και στο χρόνο αναμονής. Λέγεται ότι ε, δεν θεωρούμε όμως ότι αυτά βασίζονται σε επιστημονικές εκδόσεις, ε, ανδείξεις, συγγνώμη, δεν είναι ε, πράγματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και θα υπάρχουν ε, δραματικές συνέπειες για το πλήρωμα διότι θα κουραστεί και αυτό θα είναι σβάρος βάρος της ασφάλειάς του. Ένα βασικό θέμα με το χρόνο αναμονής και την επιφυλακή είναι τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να ε, ασκούν ε, το πλήρωμα καμπίνας και οι πιλότοι. Θα πρέπει να κοιμούνται και θα πρέπει να είναι καλύτερη ποιότητα ο ύπνο βάσει επιστημονικών ενδείξεων από τον συνήθι ύπνο. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι ει βάρο τη κρίση μα και αυτό φυσικά θα επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου και την υγεία μα. Οι έρευνε επίση έχουν καταδείξει ότι ο χρόνο επιφυλακή επηρεάζει και την ψυχική υγεία, αυξάνεται η κατάθλιψη και ε, η δουλειά μας είναι πολύ απαιτητική, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ε, έτοιμοι για δράση και να υπαχρυπνούμε, διότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πλήρωμα της καμπίνας είναι αντίστοιχο με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τη ασθενοφόρα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Και θεωρούμε ότι τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαράδεκτα, διότι δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Έξι ώρες ελεύθερου χρόνου δίνουν ευελιξία στους αεροπορικές εταιρείες. Πόση ευελιξία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε ένα κανονισμό εις βάρος της ασφάλειάς μας. Θα πρέπει να γίνει σεβαστός ο, ο κανονισμός ε, και το πλήρωμα ε, πρέπει να ξεκουράζεται καταλήλως πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεσή της και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλίσουν ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τις καλύτερες δεσμεύσεις για να υπάρχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα ασφάλειας και κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο και επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός αυτός δεν θα έχει ε, συνέπειες οι οποίες κατά την άποψή μας δεν έχουν αξιολογηθεί κατά Πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις τα στοιχεία και στις καλύτερες ρυθμιστικές ε, πρακτικές. Δεν θεωρούμε ότι βασίζονται στα καλά στοιχεία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Next is John Horn, who is the ECA. Ο John Horn από την ECA, την Ένωση των, ε, των Πιλότων, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πιλότων. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέγομαι Τζον Χόρν. Είμαι πιλότος με μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασίλειου. Πολλά χρόνια εμπειρίας. Πετάω την σειρά των ε, Airbus 320 και τα Boeing 747 για πολλά χρόνια και μικρές και μεγάλες ε, αποστάσεις. Είμαι αντιπρόσωπος των πιλότων που πετούν μέσα στην Ευρώπη και προς την Ευρώπη και από την Ευρώπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την θέση μας για αυτές τις προτάσεις σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια επί τη βάση πιλότων που έχουν εμπειρία στην πράξη. Εδώ βλέπετε λοιπόν μια εικόνα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Όταν μιλάτε για αριθμούς και στοιχεία και τεχνικά επιχειρήματα, σε τελική ανάλυση αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Έχετε δύο πιλότους οι οποίοι πετάνε ένα αεροπλάνο πολλές φορές σε κακό καιρό ή πολλές φορές με τεχνικά προβλήματα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Γιατί βρισκόμαστε εδώ. Γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σα ω δημοκρατικών εκπροσώπων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιλότοι πάντα προσπάθησαν να είναι ε, επικοδομητικοί, να έχουν τα καλύτερα, τους καλύτερους κανόνες ασφαλείας και εναρμονισμένες πρακτικέ. Αυτή η πρόταση όμω δεν φτάνει αυτό το ψηλό στάνταρ, το πρότυπο που χρειάζεται. Λαμβάνει υπόψη, δεν λαμβάνει υπόψη πολλά από τα γνωστά επιστημονικά δεδομένα. Και δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρησιμοποιήσει επιστημονικά δεδομένα για την πρόταση Κομισιόν. Ελπίζουμε ότι δεν μπορείτε να δεχτείτε αυτή την πρόταση. Αν αυτοί οι κανόνες παραβιάζουν τα επιστημονικά δεδομένα και εμπειρογνωμοσύνης, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε ασφάλεια. Εκτό αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίξει τώρα το ρόλο του και δώσει μια πολιτική κατεύθυνση για τα θέματα αυτά, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα ακολουθήσουμε το δρόμο της μικρότερης αντίστασης και της εμπορικής εκμετάλλευσης. Για να επανέλθω στο θέμα αυτό η ΆΣΑ έχει παραγνωρίσει ή δεν έχει λάβει υπόψη επιστημονικές εκθέσεις όταν δεν δίνει τις σωστές απαντήσεις για αυτήν. Η πρώτη της πρόταση δεν ελήφθη υπόψη και οι τρεις επόμενες εκθέσεις που ήταν ανεξάρτητες και αυτές παραγνωρίστηκαν. Τώρα η, το Συμβούλιο ε, Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι και η πρόταση είναι λαθασμένη και Μερικοί από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες που μελετούν την κόπωση θεωρούν ότι είναι λαθασμένη αυτή η πρόταση. Πρέπει μια πρόταση, όπως λένε και οι επιστήμονες, θα πρέπει να εμποδίζουν την διαταραχή του ύπνου, όπως όταν ξεκινάει κανείς πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ ή από πάρα πολλές πτήσεις την ίδια μέρα. Ή επίσης να υπάρχει μια επέκταση του χρόνου εργασίας όταν υπάρχει πραγματικός χρόνος ανάπαυσης στην πτήση και όχι με αυτά τα οποία αναφέρει η πρόταση. Και επομένως θέλουμε να περιορίσουμε στις 10 ώρες την βάρδια όταν οι προτάσεις επιτρέπουν και πάνω από 12 ώρες, το 12,5 ώρες. Αυτά τα νούμερα τι σημαίνουν για τον πιλότο όταν πετάει σε ένα πραγματικό κόσμο. Τι λένε οι επιστημονικές εμπειρογνώμησεις για τις νυχτερινές πτήσεις. από το, την έκθεση του ETSE και από τους επιστήμονες που μελετούν την κόπωση. Είπαν ότι δεν πρέπει ο μέγιστος χρόνος βάρδιας να ξεπερνάει τις 10 ώρες μέσα στη νύχτα. 10 ώρες μέσα στη νύχτα είναι το απόλυτο όριο για ασφαλή λειτουργία των πιλότων. Αυτό δεν αφορά μόνο την αεροπορία, αφορά και άλλες αυτό δεν σταματάει τι πτήσει, απλώς σημαίνει ότι χρειάζεται πρόσθετο προσωπικό πάνω από τι 10 ώρε. Η ΆΣΑ γνωρίζει αυτό το όριο από όλε τι μελέτε, εξακολουθεί όμω να το παραγνωρίζει. Γιατί, Γιατί δεν θα κάνει τίποτα μέχρι ότου το Κοινοβούλιο επιμείνει να τηρηθεί η δική του εντολή. Σας έχουν αναφέρει ήδη το πρόβλημα της επιφυλακής και το χρόνο που περνάει το ε, προσωπικό του πιλωτηρίου και των ε, καμπινών είναι πολύπλοκες υποτάσεις και τελικά μπορεί να καταλήξει το πλήρωμα του αεροπλάνου να προσιώσει ένα αεροπλάνο μετά από 22 ώρες εργασίας. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να έχουμε ένα όριο, μια απλή πρόταση. Το σύνολο του χρόνου πτήσης και της επιφυλακής δεν πρέπει να ξεπερνάει 18 ώρες. Δεν μπορούμε να προσγειώσουμε με ασφάλεια ένα αεροπλάνο μετά από αυτό το όριο. Οι προτάσεις απλώς δεν επιτρέπουν σε κανένα να είναι πιο ασφαλής. Θέλουν, απόλυτη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα για τις εταιρείες που θέλουν να έχουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όπως το έχει υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο. Εάν το Κοινοβούλιο δεν ζητήσει να υπάρξει ένα δεσμευτικό άρθρο που να επιτρέπει την επιλογή ασφαλεστέρων συνθήκων, θα χάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ζητούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει τα επιστημονικά δεδομένα και τα ιατρικά δεδομένα, τα οποία αυτή η πρόταση δεν τα λαμβάνει υπόψη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα, τους πιλότους από το αποτέλεσμα των πολλαπλών πτήσεων. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο 18 ώρες, 18 μετά από επιφυλακή και πτήση και πρέπει οι νυχτερινές πτήσεις να μην ξεπερνούν τις 10 ώρες. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να διαλέξουν πιο ασφαλείς ε, προδιαγραφές, αλλά αυτό δεν θα γίνει αν δεν υπάρχει μια σαφής διατύπωση σε ένα δεσμευτικό άρθρο. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει λοιπόν πραγματικότητα χωρίς τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει, έχουν ε, οι αρχέ ασφαλείας, Κάθριν Jones, εκ μέρους της ε, Βρετανικής ε, Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα για να δώσω και την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς της πτυτικής απασχόλησης. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πρόταση της Επιτροπής, Επιτροπής επομένως θα σχολιάσω μόνο την ε, γνωμοδότηση που δημοσιεύθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο. Ως ε, βασική ρυθμιστική αρχή του Βασιλείου ε, μας απασχολεί πάρα πολύ ασφάλεια και αναλαμβάνουμε τις ε, ευθύνε μας ως ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Γενικά θεωρούμε ότι το προτινόμενο πακέτο μέτρων διατηρεί τα βρετανικά πρότυπα ασφαλείας και θα τα βελτιώσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. η CIA συμμετείχε ενεργά στην ε, ομάδα διαμόρφωσης ε, πολιτικής και μας ε, επέτρεψε να εξετάσουμε την... να εξετάσουμε τη διαδικασία και να κάνουμε και τις απαραίτητες προτάσεις. Και συμφωνούμε και με τις προτάσεις που έχουν γίνει ως CAA, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας γιατί εκπροσωπήθηκαν όλοι οι μαζικοί φορείς ενδιαφερομένων και επιστημονικά στοιχεία. Έχουμε κάνει πολυάριθμες συστάσεις κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτής και ενθαρρύναμε η γνωμοδότηση της ΕΑΣΑ να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αρχική ε, πρόταση βάσει και των δικών μας ε, παρατηρήσεων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η κόπος επηρεάζεται και από πολλούς παράγοντες. Ε, μόνο και μόνο το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν μπορεί να ε, αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την κόπωση. Και τα χρονικά όρια είναι σημαντικά, αλλά και το επιχειρηματικό ε, πλαίσιο έχει πολύ σημαντική επιρροή στην συσσόρευση κόπωσης. Η γενική αποδοτικότητα οποιοδήποτε τέτοιου συστήματος για την κριτική απασχόληση θα εξαρτηθεί και από το πώς ε, συνδυάζονται όλοι αυτοί οι επιμέρους παράγοντες. Οι υφιστάμενες ε, προδιαγραφές της ε, αρχής μας δεν επηρεάζει μευτικές υποχρεώσεις για τους εμπορευομένους να έχουν συγκεκριμένη διαχείριση για την κόποση. Ε, με το προσχέδιο αυτό θα έχουμε κανόνες που βασίζονται στα αποτελέσματα και θα διαμορφώνουν σημαντικά νέα εργαλεία. Ο εμπορευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση ότι κατανοεί ε, τους κινδύνους που συνδέονται με την κόπωση στο πλαίσιο και τη λειτουργίας του. Θα πρέπει να δείχνει πώς ε, διαχειρίζεται αυτού του κινδύνου, είτε μέσω της δικής του ε, ευθύνη και του δικού του συστήματος διαχείρισης του κινδύνου, ή ε, υπό ένα σύστημα διαχείρισης του κινδύνου προκύπτει από την κόπωση. Αυτό θα επιτρέψει να μεταφέρει αυτή την επίβλεψη στο ίδιο το επιχειρησιακό πλαίσιο. Εδώ είναι οι μεγαλύτερε δυνατότητε για τη βελτίωση της ασφάλειας, κατά τη γνώμη μα. Η αρχή μας ε, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα ενδιαφέρομενα μέρη ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα θέλαμε να προταθεί ε, στον κανονισμό ο οργανισμός να πρέπει να κάνει επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των προτάσεων βάσει της συλλογής επιχειρησιακών δεδομένων και εμείς θα ακολουθήσουμε, θα φροντίσουμε να ε, τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις ο οργανισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ε, διαδικασία της συνεχούς ε, βελτίωσης βάσει και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ασφάλειας στις αερομεταφορές. Γενικά, εμείς ως ανεξάρτητη αρχή, ρυθμιστική αρχή, έχουμε συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης του πακέτου μέτρων. Θέλουμε να εφαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους αερομεταφορείς. Εκείνοι θα πρέπει να δείξουν πώς ακριβώς πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αυτές οι προτάσεις αποτελούν τμήμα μιας ε, γενικότερης διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης και θέλουμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε ενεργό συμμετέχοντα ε, στην ΕΑΣΑ για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Ευχαριστώ. Ο εμπειρογνώμονας ε, διαχείρισης ε, της ε, Γρύπνησης, ο κύριος Αλεξάνδρ Γκούντελ, ο οποίος είναι πρώην επικεφαλής της επιστημιστικής ομάδας του Ινστιτούτου της Αεροναυτικής Ιατρικής. Τέσσερα πράγματα θέλω να αναφέρω. Καταρχήν, θέλω να αναφέρω τα στοιχεία από τους εμπειρογνώμονες και επίσης τις απόψεις που έχουμε αποκομίσει από διάφορες εκθέσεις και τέλος θέλω να σταθώ στις προτάσεις και να τις αντιμετωπίσω με κριτικό τρόπο. Η συμμετοχή των επιστημόνων για τους ερευνητές του ύπνου, τους ειδικού στην κόποση, και τα λοιπά έχει γίνει σε δύο στάδια, το 2008 και το 2011. Στην πρώτη έκθεση, την έκθεση γνωστή ως ΜΕΜΠΟΥΣ, υπήρξε η συνένεση 10 επιστημόνων που αντιμετώπισαν συγκεκριμένα ερωτήματα. Η έκθεση αυτή δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν οδήγησε σε διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων και των επιστημόνων. Ένα δεύτερο βήμα ήταν μια έκταση τριών ανεξάρτητων επιστημόνων οι οποίοι απήντησαν ερωτήματα τα οποία είχαν τεθεί από την ΕΑΣΑ. Οι προσωρινές, ερωτη... οι προσωρινές εκθέσεις συζητήθηκαν από τους τρεις αυτούς επιστήμονες με τη συμβουλευτική ομάδα. Και στο τέλος η ΕΑΣΑ κατέληξε στην τελική της επιστημονική έκθεση χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη των επιστημόνων. Δεν υπήρξε επαφή μαζί τους. η ΆΣΑ ουσιαστικά παρα, ε, αγνώρισε όλες αυτές τις επιστημονικές πτυχές. Δύο βασικά προβλήματα υπάρχουν που έχουν να κάνουν με το χρόνο βάρδιας. Οι νυχτερινές πτήσεις και η κόποση. Εδώ υπάρχει μεγάλη συμφωνία των επιστημόνων ότι οι πτήσεις οι οποίες ξεκινούν αργά το βράδυ ή το πρωί οδηγούν σε υψηλό επίπεδο κόπωσης. Θα πρέπει να μειωθούν σε 10 ώρες αυτές οι ε, εκθέσεις, όπως φαίνεται και από το ε, μνημόνιο της NASA του 2011 και από το Γερμανικό Κέντρο για την Έρευνα του ύπνου. Η θέση της ΕΑΣ αυτή τη στιγμή είναι ενάντια με την άποψη των περισσότερων επιστημόνων. Η άλλη ε, πτυχή είναι μια πολύπλοκη, πολύπλοκη υπόθεση που είναι ε, η, ο χρόνος ανάπαυσης ο οποίος επεκτείνεται με τη χρήση τριών πιλότων. Με το να υπάρχουν περισσότεροι πιλότοι, τρεις ή τέσσερις, υπάρχει περισσότερη δυνατότητα χρόνου πτήσης. Αλλά ε, αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούν ε, ουσιαστικά αυτοσχέδια, κρεβάτια, κρεβάτια περιορισμένης ε, που δίνουν περιορισμένη ξεκούραση και αυτό δεν οδηγεί σε ύπνο ο οποίος είναι ανανεωτικός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία παράταση του χρόνου, πτήση, του χρόνου βάρδιας σε 14 ώρες τη νύχτα και μέχρι 16 ώρες σε άλλες περιπτώσεις. Η άποψη όμως της ΕΑΣΑ λέει 16 ώρες ανεξάρτητα από το αν αυτό γίνεται νύχτα ή ημέρα. Και εδώ δεν υπάρχει καμία επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που να το υποστηρίζει. Και η αύξηση του χρόνου αυτού που μπορεί να φτάσει το χρόνο πτήση σε 14-15 ώρες μπορεί να οδηγήσει και στο να καταργηθεί αυτή η δυνατότητα να ξεκουράζεται προσωρινά ο πιλότος σε ένα ε, κρεβάτι εκστρατείας. Έρχομαι τώρα στο θέμα της διαχείρισης του χρόνου και της κούρασης και του ελέγχου του κινδύνου. Υπάρχει μια γενική συνένεση ότι η καλύτερη διαχείριση της κόπωσης οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια και επομένως πρέπει να υπάρχει και μια εκπαίδευση των πιλότων στην καλύτερη διαχείριση της κόπωσης ως τμήμα της εκπαίδευσης ασφάλειάς τους. Και σε ορισμένε περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα μια τέτοια διαχείριση. Αντίθετα, θα πρέπει να, εμείς πιστεύουμε πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μονάχα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από τις Ευρωπαϊκές Αρχές ε, Ασφαλείας, ο Ζαν Μαρκ από την ΕΑΣΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες γενικές σκέψεις για την ασφάλεια της αεροπορίας και πιο συγκεκριμένα για τις τάσεις στην ασφάλεια της αεροπορίας. Το ποσοστό θνησιμότητας ε, στις εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη ε, διαιρείται με το 100 τα τελευταία χρόνια και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε στο 1 τρίτο του ποσοστού της ε, θνησιμότητας. Γνωρίζετε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας έχει κομβικό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας. Οι κανονισμοί της αεροπορίας τη σήμερα ημέρα είναι ασφαλείς κανονισμοί και ο ρόλος του οργανισμού είναι να τους κάνει ασφαλέστερους και βιώσιμους. Προς αυτό το στόχο λοιπόν, ποια είναι η συνέπεια της ε, κόπωσης ε, του πληρώματος. Ε, κάνοντας έρευνες ε, για τα ατυχήματα την τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκαν δύο ατυχήματα στα οποία είχαμε τρεις νεκρούς και, και στις δύο περιπτώσεις το πλήρωμα ε, εργάστηκε πέραν των νομίμων ορίων. Σε μία περίπτωση είχαμε υπέρβαση του χρόνου πτήσης κατά τρεις ώρες και την δεύτερη φορά δεν ε, έγινε σεβαστός ο ελάχιστος χρόνος ε, ανάπαυσης. Και επομένως αυτό αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες είναι βασικό στοιχείο όταν εξετάζουμε τι συνέπειε τη κόπωσης. Κάποια άλλα δυστυχήματα εκτός της Ευρώπης, για παράδειγμα το ε, ατύχημα το οποίο έγινε στις ΗΠΑ το Φεβρουάριο του 2009, καταδεικνύουν ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τους κανόνες αποτελεί κίνδυνο. Τη σήμερα ημέρα οι κανονισμοί είναι εν μέρη εναρμονισμένοι στην Ευρώπη ε, βάσει του συγκεκριμένου κανονισμού από το 2008 και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο οργανισμός ε, δεν έχουν λάβει αρνητικές ε, κριτικές για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο, ε, επειδή αναζητούμε συνεχώς ε, δυνατότητες αύξησης της ασφάλειας, εξετάσαμε κάποιες ε, απαιτήσει και έγινε μια πρόταση προς την, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή και περιλαμβάνονται πάνω από 30 βελτιώσεις. Οι επιστημονικές αποδείξεις είναι βασικές για τα στοιχεία αυτά. Μελετήσαμε πάνω από 50 επιστημονικές μελέτες και συνεργαστήκαμε με τρία ανεξάρτητα κέντρα για την ανάπτυξη του σχεδίου κανονισμού. Ε, ακολουθήσαμε τις συστάσεις των επιστημόνων. Ναι. Η συνεργασία με τους επιστήμονες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και επικοδομητική και μας οδήγησε στη μείωση ε, των νυχτερινών πτήσεων κατά 45 λεπτά, μείωση των ε, πρωινών πτήσεων πολύ νωρίς ε, κατά μία ώρα, επέκταση κατά 25, στις 25 ώρες αν ξεκινάει κάποιος νωρίς την πτήση του ή τελειώνει πολύ αργά, λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα στον ύπνο από την αλλαγή της ώρας και σε κάποιες περιπτώσεις όμως ο οργανισμός δεν ακολούθησε λέξη προς λέξη τις συστάσεις των επιστημόνων. Για παράδειγμα, οι τρεις επιστημονές μας μας πρότειναν να μειώσουμε τον χρόνο νυχτερινής ε, πτήσης στις 10 ε, ώρες. Η σύσταση αυτή έγινε επί τη βάση μιας επιστημονικής μελέτης που έγινε στη δεκαετία του 90 για τριγωνικές ε, ναυλωμένες πτήσεις μεταξύ Ινδονησίας και Σαουδικής Αραβίας στην περίοδο εχμής. Ε, κατά πρώτον λοιπόν το πεδίο αυτής της ε, ε, μελέτης είναι τόσο περιορισμένη που θεωρήθηκε ότι δεν μπορούμε να εξαγάγουμε γενικά συμπεράσματα επί τη βάση αυτής της μελέτης και μόνον. Δεύτερον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, η επιστημονική μελέτη ε, κατά βάση είναι ανταπόκριση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα και επομένως η απάντηση ε, εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από τον τρόπο με τον οποίο τίθεται το ερώτημα. Εάν λοιπόν ε, ρωτήσουμε ποιο είναι το μέγιστο όριο νυχτερινής πτήσης, η απάντηση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 10 όρια. Ώρες, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η κόποση εξαρτάται αποκλειστικώς και μόνο από την ώρα την οποία εργάζεται κάποιος. Αλλά οι επιστημονικές αποδείξεις ε, μας δείχνουν ότι δεν ισχύει μόνο αυτό. Ε, ισχύει επίσης και η εβδομαδιαία ξεκούραση, η, ε, ο χρόνος ανάπαυσης ε, για την αλλαγή της ώρας, καθώς και άλλες αρχές. Επομένως, τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε εμείς στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων ε, δεν ήταν ποια είναι η καλύτερη διάρκεια νυχτερινές πτήσεις, αλλά πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κόποση λόγω της νυχτερινής πτήσης. Και επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο μία, αλλά αρκετές επιστημονικές μελέτες, επομένως με μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μία πτήση 11 ωρών νυχτερινής πτήσης, συν επιπλέον ξεκούραση λόγω της αλλαγής της ώρας, συν επιπλέον ανάπαυση λόγω ε, πρωινής πτήσης και καθυστερημένης άφηξης, συν την εφαρμογή ε, της αρχής της διαχείρισης κινδύνου από την κόπωση, θεωρούνται ότι είναι τόσο ασφαλής όσο μία μία πτήση διάρκειας 10 ωρών. Για τον ε, ε, χρόνο επιφυλακής ε, στο σπίτι, τον κατοίκον χρόνο επιφυλακή, να, πρέπει να σα πω ότι αυτά διέπονται από εθνικού κανονισμού και όχι από ευρωπαϊκή νομοθεσία προ το παρόν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πληθώρα διατάξεων. τα όρια για την κατοίκον επιφυλακή κυμαίνονται από τις 6 στις 24 ώρες αναχώρα. Η αρχική πρόταση λοιπόν του οργανισμού ήταν 8 ώρες, δηλαδή πολύ κοντά στο κατώτατο όριο. Ε, ακούσαμε ότι 8 ώρες αναμο, αναμονής ε, με ε, 18 ώρες ε, πτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 20, ένα 24ωρο πλήρους κόπωσης. Ωστόσο, ε, το σκεπτικό και μόνον ότι η κατόκον επιφυλακή αντιστοιχεί σε χρόνο εργασίας δεν ισχύει, διότι έξι ώρες αναμονής ε, στο σπίτι του δεν σημαίνει ότι ο άλλος ε, δεν κοιμάται. Ε, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι 24 ε, ώρες αναμονής ε, κάποιος είναι 24 ώρες χωρίς, χωρίς ύπνο. Επομένως, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή για το χρόνο επιφυλακής. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσουμε τη διατύπωση, την οποία θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη στην διαδικασία επιτροπολογίας στις 23 Ιουλίου. Και η διατύπωση θα βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχής της διαχείρισης της κόπωσης Καταρχάς να υπάρχει οκτάωρη δυνατότητα ύπνου στο πλήρωμα και να υπάρχει προστασία και να μην υπάρχει άνω των 18 ώρων συνεχής εργασία. Και είμαστε της άποψης ότι βάσει αυτών των δύο αρχών η πρόταση ε, θα τύχει συνένεσης μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια για τον οργανισμό μετά την έγκριση των κανονισμών αυτών όπως ε, ακούστηκε και προηγουμένως, θα αρχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα για την εφαρμογή αυτών των νέων κανονισμών και θα γίνει μία αξιολόγηση τρία χρόνια μετά την εφαρμογή τους. Ο οργανισμός ε, θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία συλλογής δεδομένων είναι μια απαραίτητη κοινή προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο οργανισμός, τα κράτη-μέλη, αεροπορικές εταιρείες και τα συνδικάτα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, διότι ε, σήμερα περισσότερο από ποτέ η ασφάλεια μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εν τη ενώση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Κλουζό. Περνάμε τώρα στα μέλη. Κύριε Πέρκερ, Αλκαντράλ, κύριε Μάιστινγκ, Λίντεμπεργκ, Φώστερ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ζητήσει το λόγο. Άλλος κανείς. Εσείς αν θέλετε εγώ, δεν θα σας ε, αναγκάζω να μπείτε στο κατάλογο. Θέλετε, όχι. 11 ομιλητές. Δύο λεπτά ο καθένας λοιπόν. Να σας πω μόνο ότι πρόκειται για γύρω ερωτήσεων και απαντήσεων. Τονίζω ερωτήσεων. Κύριε Πέρκερ, έχετε δύο λεπτά για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μέχρι τώρα χρησιμοποίησα τον χρόνο πτήσης των πιλότων για να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ στο αεροπλάνο. Τώρα μετά από αυτά τα οποία ακούω δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι λίγο πιο άγρυπνος στο αεροπλάνο και να σκέφτομαι και κάπως ε, καλύτερα τι κάνω εκεί. Αλλά για να είμαι πια σοβαρός. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε και επίσης είχαμε επαφές ε, και εγώ και άλλοι βουλευτές με εκπροσώπους του προσωπικού, του προσωπικού. Όλοι αναφερθήκανε στα προβλήματα αυτά του χρόνου ε, εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της ε, νύχτας που λένε οι επιστήμονες πρέπει να περιοριστεί στις 10 ώρες και το συνολικό χρόνο βάρδιας συν επιφυλακής το συνολικό δηλαδή διάστημα ε, που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία χρονικά διαστήματα. Μου είπανε ότι αν εγώ ξεκινήσω πολύ νωρίς το πρωί την επιφυλακή μετά δεν έχω καμιά δυνατότητα να ξεκουραστώ, μπορεί να κάτσω πολλές ώρες επιφυλακή και μετά πρέπει να πετάξω. Αυτό στην πραγματικότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και μπορεί να φτάσει επομένω το άτρισμα της επιφυλακής και του χρόνου πτήσης σε 22 ώρες. Και αυτό ξεπερνάει πολλές φορές τα όρια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή. Το ερώτημά μου τώρα προς την Κομισιόν είναι το εξής. Πώς η Κομισιόν έχει καταλήξει σε προτάσεις όταν όλες οι μελέτες που έχουμε πάρει εμείς στα χέρια μας λένε ότι δεν πρέπει να ξεπεραστούν οι 10 ώρες τη νύχτα και ο χρόνος εργασίας, ενεργού, ενεργούς εργασίας συν ε, επιφυλακή δεν πρέπει να ξεπεράσει τις, 18, τις 16 ή 18 ώρες. Από πού λοιπόν αρίεται η Κομισιόν απόψεις οι οποίες δεν σέβονται αυτά τα όρια. Ευχαριστώ. Ερωτήματα, ερωτήματα, ερωτήματα λέει ο Μπράιν, ο κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, πράγματι εδώ πέρα δεν εκφράζουμε θέσεις, γιατί δεν υπάρχει καν πρόταση ακόμα επιτάπητος, αυτά θα έρθουν στη συνέχεια. Όμως, βάσει όλων αυτών των προσθέσεων που, υπο... μας έχει υποσχεθεί η Επιτροπή, βάσει των όσων είπε η κυρία Τσίκα, έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά. Προς τον κύριο Μπάλγουιν πρώτα ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει μια σύγχυση για τη διάκριση μεταξύ ε, ζητημάτων ασφαλείας και κοινωνικών ζητημάτων. Επιβεβαιώνεται ότι σε ό,τι αφορά τις συλλογικές ε, ε, εργασιακές συμβάσεις θα υπερβούν αυτές τις συμβάσεις λοιπόν αυτές τις διατάξεις και ότι θα διατηρηθούν τα κεκτημένα. Δεύτερον, προς τον κύριο Κουλουζό από την ΕΑΖΑ. Τονίσατε ότι ακόμα και αν συμφωνούσαμε για τους νέους ε, κανόνες, θα έρθει κατευθείαν μία φάση ε, σε βάθος ανάλυσης αυτών των κανόνων και μετά από τρία χρόνια θα έχουμε αξιολόγηση. Τι μορφή θα πάρει αυτή η αξιολόγηση. Θα πρόκειται για μια έκθεση που θα μπορούσε να εξετάσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να την αξιολογήσει. Ποια είναι η άποψή σας. Μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε σαν μακροπρόθεσμο επίπεδο την κατεύθυνση προς τον κύριο Τζόντς μετά. Δεν ε, άκουσα τόσο πολύ αυτή, κατά πόσο ε, σταθούν επιστημονικά όλες αυτές οι μελέτες που το καταξίζει. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τον ε, μέγιστο χρόνο εργασίας τη νύχτα, 10-11 ώρες, πόσες πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάισνα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ. Συγγνώμη που δεν ήρθα από την αρχή. Αλλά έχω ακούσει πολλά από αυτά τα οποία ετέθησαν. Άκουσα, θέλω να θέσω τρία ερωτήματα στην κυρία Τζόουν. Κατάλαβα καλά κυρία Τζόουν, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που προτείνεται να βελτιωθεί σε επίπεδο ε, προγραμματισμού να υπάρχει κάποια πρόνοια για περιπτώσεις που οδηγούν σε ιδιαίτερη ε, επιφόρτιση του χρόνου εργασίας. Για το θέμα, δεύτερο ερώτημα, για το θέμα της ε, διαχείρισης της κόπωσης. Μήπως αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση υποχρεωτικά και τώρα στον κύριο Κλούζο. Πιστεύετε ότι παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα ατυχήματα, αυτό θα πρέπει να μη μας οδηγήσει στο να είμαστε χαλαροί και αν έχει γίνει μια μελέτη που ασχολείται με τα θέματα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι αυτή δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί από ό,τι κατάλαβα οι μελέτες οι οποίες έχουν αναφερθεί ε, καλύπτουν ορισμένε μονάχα περιπτώσει, γιατί να μην κάνουμε μελέτες για όλες τις αεροπορικές γραμμές. Κύριε Λίχτεμπεργκερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ έχω κάποια ερωτήματα στον κύριο Κλουζό και τον κύριο Κούντουρ. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους επιστήμονες θεωρούνται από ότι ήταν υπερβολικά επιλεκτικές και κάπως δημιούργησαν μια ιδιαίτερα ροδόχρωα εικόνα, μια όχι τόσο ε, αντιπροσωπευτική εικόνα. Είναι γεγονός αυτό. Δεύτερον, ο συνδυασμός χρόνου επιφυλακής και χρόνου πτήσης. Για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα, κατά πόσο αυτό επηρεάζει τους ρυθμούς ύπνου. Και έρχομαι στο ερώτημα λοιπόν. Όταν υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά στοιχεία που λένε ότι παραγωγικά τη νύχτα πρέπει να μην περνάμε τις 10 ώρες, πώς εσείς με μία μονάχα μελέτη που έχετε αναφέρει θέλετε να είσαστε στις 11 ώρες. Αυτό θα ήθελα να το εξηγήσετε και για τον κύριο Μπόλτιν από την Κομισιόν. Τι είναι αυτή η ρήτρα που λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να... Ε, υπάρχει αυτή η ρήτα μη υπαναχώρησης. Γιατί τα κρατη δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε πιο ψηλό επίπεδο ασφάλειας και είναι υποχρεωμένα να παραμείνουν στο χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Και αυτό δεν είναι καν εκπεφρασμένο μέσα στην ε, πρόταση της Κομισιόν, αλλά είναι κάπου κρυμμένο σε αιτιολογικές σκέψεις. Επίσης, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν οι επιστημονικές μελέτες λένε και το λένε από πολλές ε, πλευρές και το ξέρουμε και από ιατρικές μελέτες ότι η νυχτερινή εργασία ουσιαστικά είναι πιο επαχθής και η νυχτερινή εργασία μαζί με χρόνο επιφυλακής δημιουργούν διαφορετική δυναμική από ότι ένας ε, κανονικός χρόνος εργασίας. Γιατί τότε δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω έχουμε στοιχεία τα οποία είναι γνωστά από όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν να κάνουν με τη νυχτερινή και ή επιφυλακή. Δύο λεπτά, κυρία Φώστα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, που ήρθαν εδώ εκπροσωπώντας ε, τον κλάδο. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις, όχι απλώς ερωτήσεις. Ε, κάποια από τα σχόλια τα θεωρώ μάλλον απογοητευτικά. Τρία χρόνια πέρασαν και οι ε, εκπρόσωποι του κλάδου συμμετείχαν σε μια επιτροπή και τώρα λένε μετά από τρία χρόνια ότι δεν ήταν κανένα εκεί. Τότε ποιε είναι οι ικανότητέ σα στη διαπραγμάτευση και τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτό το στάδιο. Ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που ε, παίζουν ακόμα. Πολλές φορές συζητάμε το ΚΑΠ 371 γιατί και εγώ ασχολήθηκα με το βρετανικό σύστημα για 25 χρόνια. και εγώ δηλαδή γνωρίζω εκ των έσω αυτά τα ζητήματα. Ε, μπορούμε λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις να πάμε στις 11 ώρες, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις πάμε στις 11, 12, 13 ώρες. Πώς θα φτάσει κάποιος στην Αυστραλία με μία μόνο ε, διακοπή. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές επιφυλάξεις. Το Πανεπιστήμιο Κραμφίλτ, Σαμρό Βασίλειο, αλλά και άλλα ε, πανεπιστήμια και ενώσει αερομεταφορών έχουν ε, πολλά επιστημονικά στοιχεία εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι πρόκειται για κάτι καινούριο. Είναι βέβαια σημαντικό να εξετάσουμε και τα νέα στοιχεία. Εγώ λοιπόν ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με τις πληροφορίες που μας έδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η Κάθριν συγκεκριμένα, και θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα σωματεία, η Ελιζαβέτα αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά στον Βασίλειο δεν υπάρχουν προβλήματα στα συνδικάτα, γιατί τους συνάντησα και αυτούς. Υπάρχουν μερικοί τομείς, όπως είναι η επιφυλακή και κάποια ακόμα, ε, που θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Αλλά δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Είναι θέμα ασφάλειας. Και ε, δεν ε, μπορεί κάποιο να είναι ξύπνιο μέσα στη μέση της νύχτας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να ρυθμίσει κάποιο το πρόγραμμα. Η διατύπωση είναι σημαντική. Συγγνώμη, Πρόεδρε, από μακρηγορώ. Ε, η διατύπωση λοιπόν είναι σημαντική. Χρειάζονται κάποιε διευκρινήσει για τα μέλη τη Επιτροπή. Θέλουμε να έχουμε μια επικοδομητική συμβόλη εδώ. Κύριε Μπάρκη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμένα με έχουν εντυπωσιάσει και ίσως ε, προβληματίσει κάποια, κάποιες δηλώσεις που άκουσα. Ίσως σε άλλα θέματα από αυτά που αναφέρει η κυρία Φώστερ για το θέμα τώρα της ε, επιφυλακής. Πώς μπορεί κανείς να κοιμάται με καταπαραγγελία, δηλαδή να χρησιμοποιεί αυτό το χρόνο για να κοιμηθεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί έχετε αναλύσει μόνο τα λίγα αυτά ατυχήματα που έχουν συμβεί και όχι τις μελέτες αυτές που έχουν γίνει, για τις οποίες αναφέρθηκε ο προηγούμενος συνάδελφος. Πώς αντιμετωπίζετε τα επιστημονικά πορίσματα ή δεν έχετε θέσει τις σωστές ερωτήσεις για να υπάρξει μια αντιπαράθεση μεταξύ των απόψεων. Όπως είπε και ο Δόκτωρ Γκίντερ, γιατί δεν έχετε λάβει υπόψη ορισμένε επιστημονικές μελέτες. Και όταν λέει η Κομισιόν ότι την ενδιαφέρει ο κοινωνικός διάλογος, εσείς δεν έχετε κάνει καμία διαβούλευση με τους εκπρόσωπους του των πληρωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός 1889 του 2006 προέβλεπε να γίνει μια ιατρική και επιστημονική αξιολόγηση για τις ε, συνθήκες εργασίας του πληρώματος καμπίνας. Σήμερα όμως αναφερθήκατε στην έκθεση Μέιμπους, μια ε, ανεξάρτητη μελέπη ε, την οποία έλαβε υπόψη τη ΣΥΑΣΑ. Εμείς ε, ως Ευρωβουλευτές μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη στο σύνολό της και κάποιες άλλες συμπληρωματικές μελέτες που έγιναν προκειμένου να μπορέσουμε πραγματικά γνωρίζοντας τι συμβαίνει να σκεφτούμε το ζήτημα και να προβλέψουμε κανόνες ε, που ε, τηρούν ε, τις απαιτήσει υγείας, ασφαλείας και είναι απαραίτητο νομίζω και τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να λάβουμε υπόψη αυτές τις τόσο σημαντικές απαιτήσει για όλους τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου, είτε είναι ε, ε, επιβάτες. Ευχαριστώ, κύριο Κράμερ, για δύο λεπτά. Μάικολ. Και πάλι έχει αποδειχθεί ότι οι φορείς σας δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν την πίεση των λόμπι. Κάθε πιλότος Όλοι οι πιλότοι έχουν παραδεχτεί ότι κάποια στιγμή έχουν κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όλη αυτή η ιστορία με την ε, εφημερία, το χρόνο επιφυλακής, έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ο χρόνος ε, επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας. Και εσείς θέλετε τώρα να έχετε τους πιλότες να είναι ξύπνοι για 22 ώρες με αυτόν τον τρόπο. Και δεν έχετε πει με ποιο τρόπο Αντιμετωπίστε τα θέματα αυτά. Φυσικά πρόκειται για τα λεφτά. Είναι φανερό. Οι αεροπορικές εταιρείες θέλουν να βγάλουν πιο πολλά λεφτά. Αλλά αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο πληρώνουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι στις αεροπορικές ε, εταιρείες με, για να καλύψουν το ΦΠΑ σε ορισμένε περιπτώσει και μιλάτε συνέχεια για ασφάλεια, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Επίση, ο αέρα στι καμπίνε των αεροσκαφών, ο οποίο είναι δηλητηριασμένο. Έχω θέσει πάρα πολλά ερωτήματα για αυτά τα θέματα. Εσεί δεν έχετε πει τίποτα, κουνά το κεφάλι σα. Ο Γερμανό Υπουργό Μεταφορών δεν είπε τίποτα για αυτά τα θέματα. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση, ούτε εσεί. Μα υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι του οποίου εσεί δεν αναφέρετε. Και έρχεστε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου η τύχη των επιβατών, δεν μπαίνει αυτό καθόλου στους υπολογισμούς σας. Μάικελ, δεν ήθελα να σας σταματήσω, αλλά υποτίθεται ότι αν αναφέρεσαι στον πρόεδρο της Επιτροπής και όχι στο υπόλοιπο κοινό της Επιτροπής. Να χαιρετήσω επίσης και μια αντιπροσωπεία από την ε, FNTR από την Γαλλική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών που είναι εδώ με την προσκλήση του κυρίου Ρικέ. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Ελπίζω ότι θα περάσετε καλά στην Επιτροπή μας σήμερα. Ο κύριος Γκρός για δύο λεπτά. Ο Μάθιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ερωτήματα. Όπως είπατε εσείς, οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν ανα πάσα στιγμή. Μόνο εισαγωγικά μία παρατήρηση γενικά για τους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα οι εμπειρογνώμονες να κάθονται στη δική μας θέση και να μπορούσαν να καταλήξουν σε μία σαφή ε, άποψη. Όταν κάποιος παρουσιάζει μόνο το άσπρο ή μόνο το μαύρο, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Το πρώτο ερώτημα. Όταν έχουμε τις μελέτες και οι μελέτες αυτές έχουν κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους που περιλαμβάνουν. Πώς μπορούμε λοιπόν από αυτές τις μελέτες που συζητάμε έχουν τις ίδιες παραμέτρους, έχουν τον ίδιο τρόπο, έχουν συγκρίνει αμνούς με ερήφια, είναι αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν με σύντομο χρονικό διάστημα, με μακρό χρονικό διάστημα, είναι συγκρίσιμα στοιχεία Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, για την ανάλυση του προβλήματος αυτού. Μπορεί κανείς να αναλύσει τα προβλήματα τα οποία προέρχονται και από το χρόνο εργασίας και την εφημερία. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αφορούσαν το χρόνο αυτό, αλλά ε, ελλειπείς ε, ή προβλήματα εφαρμογής. Και τέλος ένα πολύ απλό ερώτημα, δεν ξέρω αν αυτό έχει νόημα. Αν αύριο όλοι έχουν να κάνουν μια εργασία όπου είναι καθημερινή πραγματικότητα η κόποση, εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα ήθελε κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν θέλει κανείς να κάνει μια δουλειά που ξέρει ότι θα είναι πτώμα μετά από 12 ώρες. Μπορεί κάποιο να αντέξει 14 ώρε αν είναι ιδιαίτερα σε καλή υγεία και όχι 12, αλλά κάπου υπάρχει ένα όριο. Κύριε Σαβάλα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Μια μικρή δήλωση και μετά θα κάνω και την ερώτηση. Είναι άποψη αλλά θα τη διατυπώσω σε ερώτηση. Ο κόσμος των αεροπερικών εταιριών έχει αλλάξει πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όπως άλλαξαν και πολλοί άλλοι τομείς. Και το γεγονός είναι ότι ζούμε σε ένα στο κόσμο που λαμβάνει υπόψη τους μόνο τι είναι αποτελεσματικός προς το κόστος. Και μπορεί από πολιτική σκοπιάς να θέλω να υπερασπιστώ τον κλάδο, αλλά θα πρέπει να διατυπώσω την ερώτησή μου ως εξής. Προς την ΕΑΣΑ και τον κύριο Κλουζό. Γιατί δεν μας δίνετε κάποια επιχειρήματα εις βάθος για τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων και τις γνωμοδοτήσεις για το απλό γεγονός ότι υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορεί να αποδώσει ένας άνθρωπος. Ιδίως σε μια απαιτητική εργασία όπως η συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι είναι όνειδος το γεγονός ότι αναπόφευκτα αυτή θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ συνδικάτων και θα δραματοποιηθούν τα πράγματα γιατί για μένα στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Το μόνο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί δεν μας δίνεται καλύτερα επιχειρήματα διότι αυτό που λένε όλοι οι εμπειρογνώμονες και ισχύει αυτό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό όριο για την υπηρεσία επιφυλακής και από εκεί και πέρα τις ώρες πτήσης. Ο κύριος Λούτζας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω από μια παρατηρήση του συναδέλφου Πίρκερ, ο οποίος είπε ότι όταν ταξιδεύω, όπως μου συμβαίνει και εμένα, είτε δουλεύω είτε ξεκουράζομαι. Αλλά εγώ έμαθα και για κάποιους πιλότους, στους οποίους τους ζητούν να ε, ξεκουράζονται στη διάρκεια της πτήσης. Δηλαδή, να ε, χρησιμοποιούν την μία πτήση ως ε, κυβερνήτες του αεροσκάφους και να επιστρέφουν με την ίδια πτήση ε, σε ώρα ανάπαυσης όμως. Να χρησιμοποιούν δηλαδή τις ώρες της πτήσης ως ανάπαυση. Είναι σωστός τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος. Πρέπει να θεωρείται αυτός χρόνος ανάπαυσης. Για μένα δεν είναι αντίστοιχο του να μένει κάποιος στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει η κυρία Τζόουνς ή αν ε, σκοπιάς μπορεί να απαντήσει κάποιο από του εμπειρογνώμονε, του οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Ευχαριστώ και τέλος από πλευρά μου τρεις ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις για όλους. Η μία είναι μία απλή ερώτηση που απαιτεί ένα ναι ή ένα όχι. Η ε, ε, οι προτάσεις της ΕΑΣΑ λοιπόν που μας δόθηκαν κατά την άποψή σας είναι ε, επικίνδυνες και δεν προσδίδουν ασφάλεια. Αυτή είναι η ερώτηση. Ένα ναι ή ένα όχι εδώ. Δεύτερον, ποια εναλλακτική λύση θα θέλατε να έχετε αν σας είχα δοθεί το ελεύθερο. Το, η παλιά νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις νέες προτάσεις της ΕΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι μπορούμε είτε να ε, αποδεχτούμε είτε να απορρίψουμε την πρόταση και αν απορρίψουμε το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα εξακολουθήσει να ισχύει. Και η τρίτη ερώτηση προς την κυρία Jones, διότι δεν είμαι βέβαιος εάν η άποψη που μας παρουσιάσετε πάρα πολύ εύγλωτα από πλευρά τη CIA είναι άποψη την οποία συμμερίζονται και άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ωραία λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν με τις αεροπορικές εταιρείες και μετά τα συνδικάτα μετά η κυρία Τζόνς, μετά ο Δόκτωρ Κρούγκελ, μετά η ΑΣΑ και τέλος θα τελειώσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία λεπτά στον καθένα λοιπόν. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ο χρόνος, αλλά προσπαθήστε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στις απαντήσεις σας και να ξεκινήσω καταρχάς με τον κύριο Ντεβρόη. Τρία λεπτά για να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις. Κύριε Κόλιτσεκ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ναι, ήθελα, αλλά με παρακάμψατε. Σας παρέκαμψα. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, μπορείτε να λάβετε εσείς κύριε Κόλιτσεκ το λόγο, αλλά καλό θα ήταν να μας λέτε ότι θέλετε να μιλήσετε άλλη φορά. Έχω πάρα πολλές ικανότητες ως πρόεδρος, αλλά η τηλεπάθεια δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ αυτών. Δύο λεπτά. Δύο χέρια έχω μόνο, κύριε Πρόεδρε, τα οποία κουνάω. Την επόμενη φορά, αν θέλετε... θα μπορούσα να σηκώνω και το πόδι. Ε, τέλος πάντων, αν κάνετε κάτι το οποίο θα μου τραβήξει την προσοχή, τότε ε, μπορεί να ε, τα καταφέρετε. Αλλά το να κάθεστε εκεί αδρανείς, σίγουρα δεν έχει αποτέλεσμα. Δύο λεπτά, ένα και 44 έχετε, αλλά τέλος πάντων χάνει γενναιοδορίας ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν και επειδή υπάρχει διερμήνια θα μιλήσω τσέχικα. Δεν είμαι πιλότος, αλλά το θέμα του χρόνου επιφυλακής ε, και το κατά πόσον προσμετράται ως χρόνος εργασίας είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετά επαγγέλματα και ε, επαγγελματικούς κλάδους να ρωτήσω το εξής. Πώς αξιολογήσατε ποιο νυχτερινός χρόνος ε, θεωρείται κατάλληλο χρόνο. Εγώ έχω πετάξει πάρα πολλέ φορές και σε διάφορες ε, ζώνες ώρας και αυτό σημαίνει ότι σε 24 ώρες μπορεί να ταξιδεύει κάποιο και στη διάρκεια της ημέρας αλλά και στο βαθύ σκοτάδι. Πώς το αξιολογείτε λοιπόν αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει κάποιο συγκριτικό πίνακας των απαιτήσεων ε, των, απαιτήσεων των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας με ε, μία εβδομάδα, 30 ημέρες, ε, σύγκριση δηλαδή σε χρονικά όρια γιατί πραγματικά διαφέρουν αυτοί οι κανόνες ανά χώρα και όπως ε, σας είπα, επειδή έχω συζητήσει και διερευνήσει τα θέματα αυτά στο παρελθόν, έχω μιλήσει και με αρμόδιους ψυχολόγους, κανείς δεν ήταν σε θέση να μας πει ακριβώς ποιο διάστημα θεωρείται ασφαλής χρόνος εργασίας. Ε, ακόμα και στις οδικές μεταφορές έγινε μια προσπάθεια εισαγωγής ε, μικρών ε, ε, κυκλωμάτων τηλεόρασης για να παρακολουθούν τους οδηγούς, για να καθορίσουν σε ποια χρονική στιγμή ο οδηγός ή ο πιλότος στο πιλωτήριο είναι ήδη κουρασμένος. Έχετε εσείς τέτοια συγκριτικά στοιχεία. Ο κύριος Ντεβρό για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, αν δεν είναι ασφαλής η πρόταση της ΕΑΖΑ είναι εξαιρετικά ασφαλής ε, η πρόταση τη ΕΑΣΑ είναι η απάντηση. Είναι ασφαλέστερη σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Και λαμβάνοντα υπόψη και ότι οι αερομεταφορέ είναι πολύ ασφαλέ ε, σήμερα στην Ευρώπη, σίγουρα δεν θα μειωθεί η ασφάλεια. Έτσι απαντώ στο πρώτο σα ερώτημα. Δεύτερον, αν προτιμούμε του παλαιού ε, κανόνε ή του κανόνε ΕΑΣΑ. Βεβαίω, στο πλαίσιο της εναρμόνισης, ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμόρφωσης ενός ενιαίου συνόλου κανόνων για όλους τους ε, επιβάτες, προτιμούμε τους κανόνες ΕΑΣΑ. Βεβαίως από ε, σκοπιάς ασφάλειας μπορούμε να μείνουμε και στους παλιούς κανόνες, αλλά δεν θα είναι καλό για την εναρμόνιση των κανόνων. Θέλουμε ένα συνόλο κανόνων, γιατί οι αερομεταφορές δεν είναι πλέον εθνικές, γίνονται όλο ένα και περισσότερο ευρωπαϊκές ή και διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μόησον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, κατά πόσο η πρόταση της Άσα είναι ασφαλής. Εγώ δεν επεκτάθηκα σε αυτό γιατί ήταν δεδομένο για μένα ότι τα, το, τα αποτελέσματα της θέσης κανόνων από την ΕΑΖΑ θα είναι ασφαλής ως πρόταση. Επιβεβαιώνω, για λόγους σαφήνειας, ότι ναι, είναι ασφαλής η πρόταση, ασφαλέστερη σε σχέση με τους προηγούμενους κανόνες. Αν είχαμε δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο συνόλων κανόνων, και εμείς το εξετάζουμε επιστημονικά. Εγώ είμαι μηχανικός και όταν θέλω να παρουσιάσω κάτι, πρώτα το αναλύω. Ενημερώνομαι και συλλέγω στοιχεία πρώτη αντίδραση των μελών είναι ότι είναι κακή πρόταση, θα μας πλήξει, θα μας καταστρέψει. Ίσως υπάρχουν και αρνητικά όπως ανέφερα. Όμως, ακριβώς επειδή η πρόταση της ΕΑΖΑ είναι αποτέλεσμα τριετών διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι συνάδελφοι, συνάδελφοι εξ αριστερών μου συμμετείχαν και τα τρία αυτά χρόνια. Ναι, λέμε ότι η πρόταση ΑΣΑ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μετά από όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και μελετών επί της ασφάλειας. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω και το τρίτο ερώτημα, αλλά δεν μπορώ δυστυχώς. Όπως είπατε, δεν χρειάζεται να απαντήσετε μόνο στα δικά μου ερωτήματα, υπάρχουν πολλά που αναφέρθηκαν. Κυρία Τσίκα. Καλησπέρα σας και πάλι. Θα ήθελα να απαντήσω σύντομα, αλλά να σας πω κυρίως ότι όσον αφορά την πρόταση της ΕΑΣΑ και αν είναι ασφαλής ή όχι, έχουμε επιστήμονες εδώ που αυτοί είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν απάντηση. Όταν ε, ζήτησαν να δοθεί μια απάντηση για το σύνολο της πρότασης που έγινε από την ΕΑΣΑ, δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Το είπε και ο κύριος Γκούντερ προηγουμένως. δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς από πλευράς επιστημόνων. Δεύτερον, όταν εμείς αναφερόμαστε και στους κίνδυνους ε, σε κοινωνικό επίπεδο, αναφερόμαστε στην κόποση ως κίνδυνο, διότι είναι κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, για την υγεία μας. Εγώ είμαι αεροσυνοδός εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι τόσο αγχώδεις ρυθμοί πτήσεων μα αρρωσταίνουν και πολλές από τις ε, εταιρείες ε, χαμηλού κόστος χρησιμοποιούν και το ε, προσωπικό του πληρώματος ως μιας χρήσεως. Δηλαδή εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητές τους για ένα σύντομο διάστημα ενός έτους και στη συνέχεια ή το προσωπικό δεν τα καταφέρνει και φεύγει μόνο του ή απολύεται από την εταιρεία ε, διότι ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσει και τη δυνατότητα πτήσης. Πρέπει να είμαστε απόλυτα υγιείς για να μπορούμε να πετάμε. Και αν δεν έχουμε την υγεία μας, και αυτό είναι το αίτημά μας, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, εμείς δεν μπορείτε να μας ξεπουλάτε. Η υγεία μας είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλεια για να μπορέσουμε να λήξουμε την έξοδο κινδύνου με επιβάτες οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι πρέπει κάποιος να είναι ψυχολογικά έτοιμος και επομένως δεν μπορεί να είναι κουρασμένος. Για μένα είναι κάτι συνηθισμένο, το κάνω εδώ και 26 χρόνια και ε, εργάζομαι σε πτήσεις ε, μεγάλων αποστάσεων ε, παρεπιπτόντος. Ευχαριστώ πολύ. Λέτε ότι η πρόταση της ΕΑΣΑ είναι εγγενώς επικίνδυνη. Αυτό μας λέτε. Όχι. Ίσως ε, παρανοήθηκα. Δεν είπα αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση όμως που σας ετέθη. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Ναι, φυσικά. Την ε, πρόταση αυτή, την ερώτηση, πρέπει να την κάνετε στους επιστήμονες. Αυτή είναι η απάντησή μου. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που μπορούν να σας πούν αν η πρόταση της ΕΑΣΑ είναι ασφαλής ή όχι, εάν είναι εις βάρος της ασφάλειας. Εντάξει, δεν απαντάτε ούτως ή άλλως, κύριος Χόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα ερωτήματά σας σύντομα στο τέλος. Το πρώτο που θέλω να πω όμως είναι, ότι έχουμε κάνει σαφή τη θέση μας ε, ως ε, πιλότοι και έχουμε βασιστεί στις επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες. Έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν προσπάθειες διαπραγματεύσεων μεταξύ πληρωμάτων και εταιριών. Εμείς είπαμε δεν έχει καμιά σημασία τι λέμε εμεί, τι λέτε εσεί. Αυτό το οποίο λένε οι εμπειρογνώμονε για την ασφάλεια και την κόπωση, αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί θα βασιστούμε και δυστυχώ κανεί δεν δέχτηκε ένα εμπειρογνωμοσύνης. Απαντώντα στην ΕΑΣΑ, θα ήθελα να πω ότι οι εμπειρογνώμονε για την κόπωση αυτοί θα πρέπει να θεωρούν μια μελέτη έγκυρη ή όχι και όχι διοικητικό προσωπικό χωρίς επιστημονικά, επιστημονική γνώση. Μόνο οι επιστήμονες ξέρουν πώς μπορεί να εφαρμοστεί μια μελέτη και αν ισχύει ή όχι. Επίσης το θέμα της επιφυλακής. Είπανε πολλοί ομιλητέ ότι η επιφυλακή σημαίνει ότι μπορεί να κοιμόσαστε ως πιλότος στο σπίτι σας. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτή η περίοδος επιφυλακής είναι μια περίοδος, μια χρονική περίοδος που μπορεί να περιμένει κανείς από την αρχή αυτής της περίοδου να σας καλέσουν και μία στις δύο φορές σας καλούν. Πρέπει να είσαστε λοιπόν ξεκούραστοι και έτοιμοι για εργασία μέσα σε αυτό το διάστημα. Επομένως, αν μπορείτε να το ελέγξετε στην αρχή της περίοδου επιφυλακής, δεν ξεκουράζεστε, απλώς είσαστε ξύπνοι και έτοιμοι να πάτε στη δουλειά. Για τα ερωτήματα του Μπράιαν. Ναι, αν είναι ασφαλής οι προτάσεις της ΕΑΣΑ ξεπερνάν αυτό που λένε οι ειδικοί ότι είναι τα όρια της ανθρώπινης απόδοσης σε σχέση με την κόπωση. Γι' αυτό δεν είναι ασφαλής. Τι θα προτιμούσαν αν είχαμε διαλέξουμε μεταξύ του παλιού συστήματος και νέων προτάσεων της ΕΑΣ. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για μας. Λένε πολλοί ότι εδώ είναι μια βελτίωση σε ασφάλεια. Η Κομισιόν λέει υπάρχουν 30 βελτιώσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι η ΣΑΠΑΡΚΙΟΥ δεν είναι αυτό που ισχύει στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα, μια κουρελού από εθνικές ρυθμίσεις και συλλογικές συμφωνίες που καλύπτουν το θέμα αυτό. Σε σχέση με αυτό το εμβαλωματικό σχήμα την κουρελού είναι χειρότερες οι προτάσεις της ΕΑΣ. Μπορούν να βελτιωθούν. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ανασφαλείς αυτές οι προτάσεις. Υπάρχει πάντα δυνατότητα η Κομισιόν να κάνει προτάσεις που να αντιμετωπίσουν και τις δικές μας ανησυχίες και τις ανησυχίες των επιστημόνων. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, η πρόταση της ΕΑΣΑ θα ήταν αποδεκτή από μας. Χωρίς αυτές τις αλλαγές όμως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να μπορεί να πει όχι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή καλύτερες από το τωρινό σύστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Jones. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα στα ερωτήματά σας. Αν είναι, πιο, αν είναι εγγενώς ανασφαλής οι προτάσεις της ΕΑΣΑ, η απάντησή μου είναι όχι. Οι παλιές, ε, οι, ο παλιός κανονισμός απαρκιού ή οι νέες προτάσεις είναι καλύτερες. Εμείς προστηρίζουμε τις νέες προτάσεις, εφόσον εφαρμοστούν και σωστά βέβαια, και αν η άποψή μας είναι μια άποψη που είναι γενικά αποδεκτή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και θα ψηφίσουν στο Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Επομένως δεν μπορώ να απαντήσω στη θέση τους, αλλά κατανοώ από αυτά που ξέρω εγώ ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τις νέες προτάσεις όσες έχουν. Αλλά φυσικά δεν μπορώ εγώ να πάρω τη θέση των κρατών μελών. Τώρα είναι πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Προσπαθώ να θυμηθώ λιγάκι. για τα όρια της νυχτερινής εργασίας. Πολλοί συζητήσανε τι θα πει νύχτα. Αυτό είναι μεταξύ των 2 και των 4.59 το πρωί, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Οι προτάσεις που αναφέρονται θα επικαλύπτονται κατά μία ώρα και 50 λεπτά στον χρόνο. Θα μειώσουν μάλλον το χρόνο που θεωρείται νυχτερινό για μία ώρα και 50, Επίση αυτό θεωρούμε ότι είναι στοιχείο ασφαλεία. Επίση θεωρούμε ότι η πρόταση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικέ αρχές. Μία από τι βασικές επιστημονικέ αρχές είναι ότι το όριο χρόνου είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εργασίε που γίνονται πριν και μετά και ο χρόνο ανάπαυση που είναι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει η σωστή διαχείριση του χρόνου εργασίας πέραν από τις 10 ώρες, οι δικές μας έρευνες και τώρα και σε ιστορικό επίπεδο δείχνουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και πέρα από τις 10 ώρες. Αλλά οι νέοι κανόνες λένε ότι πρέπει να υπάρχει ενεργή, διαχείριση του πρόσθετου αυτού χρόνου και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι περιορίζει το επίπεδο ασφαλείας. Για τα ημερήσια όρια. Από την πλευρά της ασφάλειας θα πρέπει να δούμε πότε πετάει το αεροπλάνο το πλήρωμα. Επομένως δεν θα θέσουμε ε, ημερήσιο όριο, κοιτάμε απλώς το χρόνο πτήσης. Οπότε θα είναι δυνατό για ένα μέλος του πληρώματος μετά από ε, το χρόνο πτήσης να ξεκουράζεται και αν είναι 24 ώρες το χρόνο εργασίας θα πρέπει να έχουν 24 ώρες ε, ανάπαυσης. Νομίζω ότι αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Γούντελ. Τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον έλεγχο ε, ε, τη διαχείριση της κόπωσης, αν γίνεται σωστά, συμφωνώ ότι μειώνει τους κινδύνους. Το δεύτερο έχει να κάνει με, την, ε, με το πόσο ειδικέ είναι οι ερωτήσεις της ΕΑΣΑ για τις μελέτες αυτές. Μπορείτε να τις βρείτε λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά μπορεί κανείς να πει γιατί αυτές οι ερωτήσεις και όχι άλλες ερωτήσεις αλλά νομίζω σε τελική ανάλυση αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή είναι η απόψή μου τουλάχιστον. Ο κύριος Γκρός θέλει να ξέρει πώς μπορεί κανείς να συγκρίνει τις μελέτες και το, οι μελέτες αυτές που είναι το 89 και το 95 υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, ε, Ιαπωνίας, Ευρώπης και ήμασταν ομόφωνοι, όπως και το 89, ότι πρέπει να περιοριστεί ο χρόνος νυχτερινής ε, πτήσης σε 10 ώρες. Και έγιναν μελέτες οι οποίες έγιναν από την ΆΣΑ, οι οποίες όμως δεν θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα έγκυρες. Το θέμα της επιφυλακής. οι πιλότοι πρέπει όταν θεωρούν ότι δεν είναι έτοιμοι να πετάξουν να πούν ότι είναι κουρασμένοι και δεν μπορούν να πετάξουν ακόμα και μετά από ένα χρόνο επιφυλακής. Και υπήρξε το ερώτημα στα Ιταλικά από τον κύριο Γκίας για τον χρόνο ε, ανάπαυσης, για τον χρόνο επιφυλακής. Αλλά ο χρόνος επιφυλακής δεν μπορεί να είναι χρόνος ανάπαυσης, είναι χρόνος εργασίας. Τα ερωτήματα τώρα του Πρόεδρου. Εγώ δεν μπορώ τώρα να δώσω μία ε, απάντηση η οποία θα τρομοκρατήσει ένα τμήμα του πληθυσμού. Γενικά έχουμε αν έχουμε προτιμούμε τους κανόνες της ΕΑΣΑ ναι εάν υπάρξουν και ενσωματωθούν οι προτάσεις βελτίωσης που ε, λέγονται δεσμένοι θα είναι καλύτερες. Δεν μπορώ από τώρα ότι είναι καλύτερες από αυτό που έχουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Κλουζά, έχετε τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στα επιστημονικά ζητήματα και ελπίζω μαζί με τον Ματιού να καταλήψουμε όλα τα ερωτήματα. Για την επιστημονική μελέτη που θα εκπονήσει ο οργανισμός ε, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή των κανόνων. Ο οργανισμός ε, θα δημοσιεύσει λοιπόν μια έκθεση μετά από αυτή την ε, μελέτη και αυτή η έκθεση θα δημοσιευθεί και στον ιστότοπο της ΕΑΣ, θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό διαθέσιμη η έκθεση στο ευρύ Και προς τα μέλη του Κοινοβουλίου βεβαίω ε, θα απευθύνεται και με τα χαρά να τη συζητήσουμε. Μετά, εάν δούμε ότι μένουν ακόμα να επέλθουν κάποιες ε, βελτιώσεις ό,τι αφορά την ασφάλεια, σίγουρα και μπορούμε να τι κάνουμε. Ε, αναφέρθηκε η μείωση των ατυχημάτων. Όμως, όπως σας λέω, ότι μειώθηκε το ποσοστό των ατυχημάτων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς σταματούμε να προαγάγουμε την ε, βελτίωση του επίπεδου ασφαλείας. Αντιθέτως, μετά αναφέρθηκε ότι κατά πόσο ε, μας επηρεάζει το πού γίνονται οι μελέτες. Πράγματι, γιατί στις ΙΠΑ μπορούν να έχουμε 14 ώρες ε, ε, απασχόληση και 10 ώρες ανάπαυσης, ενώ εδώ έχουμε 14 ώρες ε, εργασίας και 18 ώρες ανάπαυσης. Επομένως, στις ΕΙΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερη κόποση. Επομένως, αν συγκρίνεται τα αποτελέσματα αντίστοιχων μελετών, είναι εντελώς διαφορετικά στις ΕΙΠΑ και στην Ευρώπη. Για την έκθεση Μόιμπους, την οποία έχει δημοσιεύσει ο οργανισμός τον Ιανουάριο του 2009 και γιατί δεν ε, τηρήσαμε απόλυτα αυτά που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση. Δεν ξέρω αν εδώ θα είναι πολιτικά ως ορθό αυτό που θα σας πω, αλλά δεν ήταν καλή αυτή η έκθεση σε όλες τις περιπτώσεις. Και ενέκρινε μελέτη που έγινε στη ΣΥΠΑ από στατιστικολόγο που δεν έχει καμία επιστημονική γνώση για τα ζητήματα που αφορούν τις αερομεταφορές. γιατί δεν ε, ακολουθήσαμε και δεν ε, λάβαμε τη σύμφωνη γνώμη των επιστημόνων. Αυτό συνέβη. Είχαμε συνεδριάσεις με τους επιστήμονες, τριήμερες και συνεχείς επαφές με τους επιστήμονες κατά την εκπόνηση της έκθεσης και θεωρούμε ότι έτσι έχουμε επαρκή συμβολή από τον επιστημονικό κλάδο. Αυτά είχα να προς το παρόν. Κύριε Μπόλτουιν, Μάικλ, συγγνώμη. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί. Κύριε Μπόλτουιν, τους δίνουμε μόνο τρία λεπτά έτσι κι αλλιώς. Κατανοείτε λοιπόν. Κύριε Μπόλτουιν, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κι εγώ όσο μπορώ περισσότερες ερωτήσεις μέσα στα τρία λεπτά που μου δίνετε. Αναφέρθηκαν πολύ σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την επιφυλακή και εκτός αεροδρομίου μάλιστα. Το θέμα είναι εάν η γνωμοδότηση ΆΣΑ και αν οι προτάσει τη επιτροπή θα επιτρέψουν σε μία ασφαλή, σε, πρότυπα. Η απάντηση είναι όχι. Για δύο κύριους ε, λόγους. Πρώτον, συγγνώμη, προσπαθώ να απαντήσω. Πρώτον, επειδή η πρόταση της ΆΣΑ ε, θέτει ρητός υποχρεώσεις προς κράτη-μέλη, αερομεταφορές και προσωπικό ότι διασφαλίζουν ε, την, ε, τον έλεγχο της εκόπωσης. Αυτές οι διατάξεις ε, υπερέχουν των μέγιστων ορίων και πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί, πρέπει όμως να σκεφτόμαστε ότι και οι εθνικές αρχές ελέγχουν την, τις διατάξεις ασφαλείας. Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να αξιοποιεί και τη δυνατότητα ανάπαυσης κατά τη διάρκεια επιφυλακής, γιατί γνωρίζουν και ποια είναι τα, ποιες είναι οι ώρες εργασίας τους. Ε, μετά, το προσωπικό δεν είναι αναγκασμένο να εργαστεί όταν θεωρεί ότι ε, τελεί υποπερκόπωση. Μετά αναφέρθηκε ότι μπορεί κάποιος να μείνει εξύπνιος 24 ώρες. Αυτό είναι λάθος. Αν δεν τον καλέσει η αεροπορική εταιρεία, τότε θα μείνει στο κρεβάτι του βεβαίως. Και δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να σηκωθεί ο άνθρωπος να φτάσει στη δουλειά του. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε πάνω από 18 ώρε ε, να είναι κάποιος ξύπνιο. Αυτό είναι λογικό βάσει των επιστημονικών μελετών. Κάτι άλλο αφορούσε τι νεκτερινές πτήσει. Εδώ πράγματι αναγνωρίζω και σέβομαι μετά όσα αναφέρθηκαν. Ξέρετε ότι δεν επιτρέπουμε 11 ώρες και 45 λεπτά νυχτερινής πτήσης. Οι, τα, οι προτάσεις σε άσα θα προστατεύουν ακόμα περισσότερο προσωπικό, έχουν 4 μέτρα, μειώνουμε το όριο στις 11 ώρες Δεύτερον, καλούμε τους εμπορευομένους να ε, εφαρμόσουν προγράμματα διαχείρισης ε, κόπωσης για πάνω από τις 10 ε, ώρες κατά τη νύχτα και ζητούν και επιπρόσθετους, επιπρόσθετη ανάπαυση εβδομαδιαίως 60 ώρων αντί για 36 σε περίπτωση διαταραχής του ύπνου. Μετά, σύνδεση κανόνων ασφαλεία και κοινωνικών ε, ε, ζητημάτων. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα επιτρέψουν την εφαρμογή ε, προστατευτικών μέτρων στι συλλογικέ συμβάσει. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του συστήματος πτυτική απασχόληση και των διαπραγματεύσεων στις συλλογικές συμβάσει. η σύνδεση μεταξύ των δύο λοιπόν βασίζονται στην αρχή ότι ισχύει ο πιο προστατευτικό κανόνα οι διατάξεις του νέου κανονισμού βεβαίως ε, εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη της εθνική νομοθεσία και των ε, συλλογικών συμβάσεων εργασία. Κυρία Λίχτεμπερ και άλλοι ρώτησαν αν το κράτος μέλος θα μπορέσει να εφαρμόσει πιο ε, προστατευτικά μέτρα από ότι οι κανόνε ΕΑΣΑ. Πράγματι, βάσει του κανονισμού, οι εναρμονισμένοι κανόνε ασφαλεία αντικαθιστούν τους εθνικούς κανόνες για να υπάρχει ένα καλύτερο ισότιμο πεδίο δράσης. Όμως, ε, οι εθνικές ε, παρεκκλήσεις ε, μπορούν να εφαρμόζονται αν όμως υπάρχει κοινοποίηση προς την ΕΑΣΑ. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες μεταξύ χωρών για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία όπου υπάρχουν περίοδοι ε, όπου η νύχτα είναι μεγάλη. Δεν θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει μια νέα διάταξη που να διευκρινίζει ότι μπορούν να υπάρξουν παρεκκλήσεις, γιατί οι φυστάμενοι κανόνες είναι ξεκάθαροι κατά τη γνώμη μας. όλα αυτά, είμαστε διατεθειμένοι να το εισαγάγουμε αυτό σε μια αιτιολογική σκέψη. Να απαντήσω τώρα στον κύριο Κρέμερ για ε, το πλήρωμα ε, θαλάμου, ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εμείς, ε, αυτοί οι κανόνες ισχύουν και για τους πιλότους και για το πλήρωμα του θαλάμου. Και στην πρότασή μας αυτή και στη συνεργασία μας με τα συνδικάτα, ε, και λυπάμαι που κάποιοι δεν το αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά μας, σε ό,τι αφορά την ανάπαυση εντός του αεροσκάφους για το πλήρωμα, η ΆΣΑ θα προτείνει μια τροποποίηση, μια προσαρμογή που θα διευκρινίσει κάτι που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τη συζήτηση με τα σωματεία. Δυστυχώς δεν έχω παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Baldwin. Κάποια τελικά σχόλια από μένα και από τον κύριο Αλκουαντράουι, ο οποίος είναι ειδικός για τα θέματα επιτροπολογίας. Θες να πεις κάτι, Σαΐντ. Μπράιαν, δεν χρειάζομαι 50, 15 λεπτά. Για μένα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν βέβαια όλοι. Μας βοηθάει όμως να καταλάβουμε καλύτερα τι διακυβεύεται και ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Κάποια στιγμή πριν από το καλοκαίρι η Κομισιόν θα πρέπει να οριστικοποιήσει την πρότασή της και από ό,τι ακούω μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις οι οποίες είναι υποσυζήτηση από τους εμπλεκόμενους και πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες έχει βοηθήσει για να έλθουν πιο κοντά οι εμπλεκόμενοι. Γιατί πράγματι θα προτιμούσαμε να έχουμε κάτι το οποίο είναι γενικά αποδεκτό από όλους. Και ελπίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι όταν υπάρχει η οριστικοποιημένη πρόταση θα μπορέσουν να απαντήσουν στο ερώτημά σας που είναι αν προτιμάτε την τωρινή πρόταση ή την προηγούμενη αν θεωρείτε ότι υπάρχει βελτίωση σε ασφάλεια ή όχι. Και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι μπορούμε απλώς να δεχτούμε ή να απορρίψουμε την πρόταση ως σύνολο και έτσι να σπαταλήσουμε τα τρία χρόνια προπαρασκευαστικής εργασίας που έχουν λάβει χώρο. Αυτή η απόφαση λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ καλά σταθμισμένη. Ευχαριστώ. Και από μένα κλείνοντας. Να σας υπενθυμίσω ότι εγώ ήμουνα ο εισηγητή για το πακέτο EU Ops στο παρελθόν. Ακόμα έχω τις ουλές από αυτή τη διαδικασία που χρειάστηκε ένα απίστευτο χρονικό διάστημα για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία για να μπορέσουν και οι κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν. Από κάποια άποψη η παλιά ρύθμιση είναι δικό μου μωρό. Έχει τη σφραγίδα του Brian Simpson. Μέσα στο πλαίσιο αυτό όμως πάντα θα πρέπει να την χάνει αναθεώρησης και βελτίωσης και αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα αυτό. Τι προτιμάτε την παλιά ρύθμιση ή την τωρινή ρύθμιση που προτείνεται. Γιατί δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι θέλουμε λίγο από αυτό και λίγο από εκείνο. Ή το παλιό ή το καινούριο θα επικρατήσει. Αυτή είναι η επιλογή λοιπόν, που έχει το Κοινοβούλιο. Όταν τελικά υποβληθεί η πρόταση Κομισιόν και καταλαβαίνω πόσο η επιλογη που εχει το κοινοβουλιο είναι αυτό για όλους μας γιατί είμαστε στο σκοτάδι, γιατί φανταζόμαστε πώς θα είναι η τελική πρόταση της Κομισιόν, αλλά επισήμως δεν έχουμε ακόμα τίποτα στο οποίο να βασιστούμε. Τούτου λεχθέντος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή την ε, μήνυα ακρόαση. Τον κύριο Μπόλτουιν, τον κύριο Ντεβεράη, Μόισεν, την κυρία Τσίτσα, τον κύριο Χολ, Jones, τον Δόκτωρα Γκούντουλ και τον Δόκτωρα Κλουζό. Και ευχαριστώ όλα τα μέλη που έμειναν εδώ. Μόνο σε ένα σημείο κάπως διαταράχτηκε η πειθαρχία της Επιτροπής, αλλά γενικά ήταν πολύ καλή και υπήρξαν πολύ ενδιαφέροντα και εύστοχα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει η πρόταση της Κομισιόν και θα δούμε τι θα προκύψει. Τώρα συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας και κλεισμένων των θυρών. Δύο-τρία λεπτά διακοπή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και κλεισμένων.